Here we go. All right, welcome everybody. Uh, ορίσατε, συνάδελφοι. Ο πρόεδρος Μπούζεκ θα έρθει σε μια ωρίτσα. Στο μεταξύ έχω το προνόμιο να προεδρεύω εγώ σε αυτή τη συνεδρίαση. Καταρχάς ε, πρέπει να εγκρίνουμε πρακτικά συνεδριάσεων από τον Ιούλιο ακόμα. Αν δεν υπάρχουν λοιπόν ε, ενστάσεις μέχρι το πέρας της σημερινής συνεδρίασης, ε, θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά να περάσουμε τώρα στο προκείμενο, στο εργαστήριο για το Brexit και τη βιομηχανία και την ε, πολιτική διαστήματος. Να καλωσορίσω όλους τους συμμετέχοντες. Πρόκειται για το τρίτο εργαστήριο, σε μια σειρά εργαστηρίων που κάνουμε για τις συνέπειες του Brexit και την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27 και έχουμε ένα τελευταίο για το Brexit και τον, ε, το Horizon Europe που θα γίνει τον Νοέμβριο. Η βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει στόχο να κάνει την ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανταγωνιστική, ώστε να διατηρήσει το ρόλο της ως μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης και απασχόλησης στην Ευρώπη. Οι πολύ μικρέ και μικρομεσαίες επιχειρήσει αποτελούν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παρέχουν τα 2 τρίτα των θέσεων εργασία του ιδιωτικού τομέα και συμβάλλουν σε περισσότερο από το ίμιση της περιοριστηθάμενη αξία που δημιουργείται από τι επιχειρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια ισχυρή πολιτική διαστήματο μπορεί να ωφελήσει και την επιστημονική έρευνα, αλλά και την ευρωπαϊκή οικονομία εν γέννη, καθώς επίση σε τομεί όπω είναι οι μεταφορέ και το κλίμα, αλλά και επικοινωνίε και ασφάλεια. Μας μένει λιγότερο από ένα εξάμεινο μέχρι το Brexit και στο σημερινό εργαστήριο θα εξετάσουμε τις πιθανές νομικές και οικονομικές συνέπειες της Ευρώπης των 27, ε, του Brexit για τη βιομηχανία και την ε, πολιτική διαστήματος. Είναι αναπόφευκτο να μην υπάρξει κάποιος αντίκτυπος από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Έχουμε κάτι λιγότερο από μια ώρα, γιατί θα ψηφίσουμε στις 4 η ώρα. Το εργαστήριο μεταδίδεται ζωντανά στο διαδίκτυο. Θα αναρτηθούν ε, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ήτρε και οι παρουσιάσεις. Θα υπάρχει και μια συνοπτική έκθεση και οι ομιλητές θα έχουν το πολύ 10 λεπτά αναπαρουσίαση. Μετά από την παρουσίαση των τριών ομιλητών μας ε, θα έχουμε και ε, δυνατότητα για ερωτήσεις και απαντήσεις. Να δώσω λοιπόν το λόγο στον πρώτο ομιλητή, η Ράιν Χίλντε Βόγγελερ, δεν ξέρω αν πρόφερα σωστά το όνομά σας, η οποία θα μας παρουσιάσει μια εικόνα των πιθανών επιπτώσεων ε, του Brexit ε, για την βιομηχανική πολιτική και την πολιτική διαστήματος της Ευρώπη των 27. Η κυρία Βόγγελερ είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο KU11, στο τμήμα διαχείρισης στρατηγικής και Κοινοτομίας. είναι ε, μέλος του Μπρούγκελ από το 2009, είναι επίσης ερευνητικός ε, ε ερευνήτρια μάλλον, συγγνώμη, στο CRP και μέλος της ε, ε, Βασιλικής ε, Φλαμαδικής Ακαδημίας του Βελγίου και Επιστημών. Αυτή τη στιγμή είναι και επιστημονική σύμβολος και μέλος του ε, Τμήματος Πολιτικής του Επιτρέπου Κάρλος Μόετας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα να μιλήσω για τη βιομηχανία και την πολιτική διαστήματος και πώς θα διαμορφωθεί μετά από το Brexit. Το πρώτο σημείο με το οποίο ξεκινούν όλες οι εκδηλώσεις για τον Brexit είναι ε, πώς ε, θα διαμορφωθούν οι εμπορικές σχέσεις ε, μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27 και βεβαίως υπάρχει όλη η βεβαιότητα για το πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα μετά τον Brexit, τι στρατηγική διαστήματος θα αναπτύξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο βεβαίως αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση να εξετάσει πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί η βιομηχανική πολιτική και η πολιτική διαστήματος ε, αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα λοιπόν. Εδώ μπορούμε να αναφέρουμε μόνο κάποιες γενικές αρχές για τον τρόπο με τον οποίο θα απαντήσει η βιομηχανική πολιτική και η πολιτική διαστήματος των 27 και αυτό θα προσπαθήσω να κάνω εδώ στην παρουσίαση. Θα έχουμε μια ευρεία παρουσίαση των αρχών αυτής της ε, πολιτικής ε, και σε βιομηχανικό επίπεδο και σε επίπεδο διαστήματο και οι άλλοι δύο μιλητέ ε, θα επισέλθουν σε πολλέ λεπτομέρειε για τη βιομηχανική πολιτική και την πολιτική διαστήματο. Εγώ θα σα παρουσιάσω ένα σκαρίφωμα λοιπόν για το τι γίνεται και ποιο είναι ο αντίκτυπο και πώ μπορούμε να κατανοήσουμε το γεγονό ότι αλλάζει αυτό το περιβάλλον και να δούμε και τι πολιτικέ θα χρειαστούμε ε, στην Ευρώπη των 27 για να υπάρξει ανάπτυξη τι είδους πολιτική λοιπόν θα χρειαστούμε σε θέματα βιομηχανίας και διαστήματος και μετά θα δούμε και τι αντίκτυπο θα έχει το Brexit για αυτές τις απαιτούμενες πολιτικές. Όσον αφορά τις προκλήσεις και τις αλλαγές στο περιβάλλον, Νομίζω ότι περισσότεροι είστε εξοικειωμένοι από αυτά. Αυξάνεται η παγκοσμιοποίηση, ιδίω αναδύονται χώρε όπω η Κίνα ε, η Ασία εν γέννη. Επίσης, ψηφιακές τεχνολογίες, οι οποίες εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα και κατά συνέπεια υπάρχουν και πάρα πολύ ε, θολά όρια μεταξύ διαφέρων ε, τομέων. Για παράδειγμα, ε, έχουμε πλέον υπηρεσίες στην μεταποίηση. Είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε σαφή διάκριση μεταξύ των διαφέρων τομέων λοιπόν και φυσικά αυτό σημαίνει ότι είναι θολά και τα στενά όρια και έχουμε περισσότερα πράγματα που οποία συνδύονται με παγκόσμιες αλυσίδες αξιών. Και φυσικά αυτά επηρεάζουν και το περιβάλλον για τις επιχειρήσεις ε, που είναι εκτεθειμένες πλέον σε πολύ περισσότερη αβεβαιότητα και οικονομική, αλλά και πολιτική με την αύξηση του προστατευτισμού των εμπορικών πολέμων και το Brexit φυσικά, που είναι στοιχείο αβεβαιότητας, αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο. Πολύ μεγαλύτερη αβεβαιότητα λοιπόν σε σχέση με την πολιτική εγγένεια να σας πω ποιος είναι ο πολύ σημαντικός ε, μοχλός των αλλαγών που θα συζητήσουμε. Αυτή η τάση για την παγκόσμια λυσίδα αξιών και τη σημασία της δυνατότητας καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερευνήσαμε λίγο το θέμα στον Μπρούγελ για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε τα καλύτερα στοιχεία και βλέπουμε ότι οι οικονομικές δραστηριότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ καλύτερα ενσωματημένε ε, στι παγκόσμιες ε, αλυσίδες αξιών και φυσικά έχουμε και αυξημένη εξειδίκευση, όχι στον τομέα απαραίτητα, αλλά σε συγκεκριμένα ε, στάδια και καθήκοντα εντός τη αλυσίδα. Και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ε, κοινή σχέση και δημιουργείται αξία ε, σε επιχειρήσεις, σε ενδιαφέρου κλάδους και μεταξύ χωρών. Επίσης διαπιστώνουμε από τα στοιχεία που έχουμε ότι παρά το γεγονός ότι συνήθως χρησιμοποιούμε τον όρο παγκόσμια αλυσίδα αξιών. Ε, υπάρχει για την Ευρώπη μια ευρωπαϊκή διάσταση πολύ σαφής και πολύ συχνά οργανώνονται σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο αυτές ε, οι αλυσίδες. Επομένως μπορούμε να μιλήσουμε για ευρωπαϊκές αλυσίδες αξιών. Αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτές τις αλυσίδες αξιών και δεν είναι μόνο οι μεγάλες επιχειρήσεις που βρίσκονται επικεφαλής, αλλά και μικρομισές επιχειρήσεις, μικρές επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες ε, σε αυτές τις επιχειρήσεις μπορεί να επιτύχουν πολύ πιο βιώσιμες αντικανονιστικές θέσεις, θα είναι πολύ πιο παραγωγικές και φυσικά θα έχουν περισσότερη αξία και φυσικά εάν η συμβολή τους βασίζεται σε μοναδικές δεξιότητες και προσόντα, ε, όταν θα ευθυγραμμιστούν στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξιών θα έχουν πολύ μεγαλύτερη αξία. Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα καινοτομία και στις παγκόσμιες αλυσίδες αξιών γιατί έτσι θα μπορούμε να βασιζόμαστε σε επιχειρήσεις και σε διαφέρους κλάδους για να συμβάλλουν στην ευρωπαϊκή οικονομία όχι τόσο όσον αφορά την ποσότητα που παράγεται, αλλά περισσότερο ε, την ποιότητα των όσων παράγονται και έτσι θα μπορέσουν να συμβάλλουν με αύξηση παραγωγικότητας και ε, δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενες αξίες, οι οποίες πολύ συχνά ε, συνδέονται και με τη δυνατότητα καινοτομία. Και αυτό φυσικά το βλέπουμε σε όλους τους τομείς ε, και επομένως η συμβολή έρχεται από δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενες αξίες, οι οποίες βασίζονται σε δυνατότητες καινοτομία επιχειρήσεων που σχεδιάζουν αυτέ τι δυνατότητε και αυτέ τι δραστηριότητε εντό ε, παγκοσμίων αλυσίδων αξιών και στην Ευρώπη ευρωπαϊκών αλυσίδων. Πώς μπορούμε εδώ να σχεδιάσουμε την πολιτική μας. Πρέπει να δούμε ότι είναι συνδεδεμένες αυτές οι δραστηριότητες και μεταξύ επιχειρήσεων και μεταξύ κλάδων αλλά και μεταξύ χωρών. Και επίση θα πρέπει να δούμε και ε, τι συνέπειε υπάρχουν για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να σχεδιάζονται οι πολιτικέ. Ε, δεν θα πρέπει να υπάρχουν μόνο αυτέ οι αλυσίδε, αλλά να μπορεί κάποιο να υποφελείται και τη αλυσίδα. Που σημαίνει ότι σε πρώτο βαθμό πρέπει οι αλυσίδε αυτέ να μπορούν να δραστηριοποιούνται. Διασυνοριακέ ροέ κεφαλαίων, ανθρωπίνου δυναμικού και γνώσεων φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικά αλλά επίσης είναι σημαντικό να υπάρξει και αξία βάση αυτών. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι κάθε χώρα θα πρέπει να τα συνδάσει αυτά με δυνατότητες παραγωγικότητας σε καθήκοντα επί των οποίων θα εξειδικεύονται σε αυτές τις παγκόσμιες αλυσίδες. Χρειαζόμαστε λοιπόν ρευστές αλυσίδες αξιών και οι χώρες ε, θα πρέπει να εξειδικεύονται όμως και ε, να ενσωματώνουν κάποια καθήκοντα που ε, ε, διαθέτουν σε τοπικό επίπεδο εντός της αλυσίδας. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε πάντα ένα συνδυασμό εμπορικών πολιτικών, πολιτικών συνόρων δηλαδή, για να διασφαλίσουμε την καλή λειτουργία αυτών των αλυσίδων αξιών, αλλά για να μπορέσει κανείς να ε, έχει αξία, θα πρέπει να δει και τι γίνεται πέραν των πολιτικών των συνόρων, να μπορεί να έχει συμμετοχή και αυτό είναι σημαντική, λοιπόν, ε, σημαντικό γιατί έχουμε συνδυασμό της εμπορικής πολιτικής ε, και της πολιτικής που διέπει όλες τα υπόλοιπα πράγματα εκτός των συνόρων. Θα πρέπει λοιπόν να μπορούμε να ε, εντάξουμε ε, όλες αυτές τις δυνατότητες με ανοιχτό πνεύμα σε ε, διεθνή ε, δίκτυα παραγωγής και φυσικά να έχουμε τις αλυσίδες. Αυτό σημαίνει καταρχάς ότι για να μπορέσουμε να έχουμε αξία από αυτές τις ευρωπαϊκές ε, αλυσίδες αξιών. Θα πρέπει να έχουμε ευρωπαϊκές πολιτικές ε, εμπορίου και φυσικά δασμολογική και μη δασμολογική φραγμή επειδή ε, μεγιστοποιούνται, ε, εάν υπάρξουν σε οποιοδήποτε σημείο θα έχουν πολύ μεγαλύτερε συνέπειε σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανοιχτέ αγορέ ε, και άρση εμπορικών και δασμολογικών και μη δασμολογικών φραγμών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό σημαίνει ότι όλε οι συνιστώσει τη αλυσίδα αξιών πρέπει να είναι αρκετά ανοιχτέ, αλλά επίση θα πρέπει να σκεφτόμαστε και ευρύτερα όσον αφορά του εμπορικού μα εταίρου. Διότι οποιοδήποτε πρόσκομα που υπάρχει με τρίτη χώρα που συνδέεται με κάποιο τρόπο με την αλυσίδα θα έχει συνέπειες για όλους. Και αυτό δεν είναι μόνο προς την ε, ε, άμεση κατεύθυνση, αλλά και για άμεσους, έμεσους εταίρους. Η απελευθέρωση λοιπόν του εμπορίου θα πρέπει όλο ένα και περισσότερο να γίνει περισσότερο πολυμερής για να μπορέσει να ε, δει και τις άμεσες αλλά και τις έμεσες συνέπειες. Και φυσικά δεν αφορά μόνο ε, φραγμούς, αλλά υπάρχουν και θέματα προτύπων, παραγωγής και προδιαγραφών και αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Η νέα αγορά λοιπόν είναι πολύ σημαντική. Επίσης, αυτοί που προμηθεύουν με ε, ανταλλακτικά και εξαρτήματα θα είναι πολύ σημαντικοί εδώ και θα πρέπει φυσικά να είναι επαρκώς οικονομική σύνδεση. Χρειαζόμαστε λοιπόν παγκόσμια δίκτυα παραγωγής ε, και κατάλληλες αλυσίδες επιμελητίες. Να υπάρχουν λοιπόν κατάλληλες υποδομές και συμπληρωματικές υπηρεσίες που να είναι επαρκώς ε, ενταχμένες για να μπορέσουμε να έχουμε και τοπική ε, ένταξη. Πρέπει λοιπόν να έχουμε όλες αυτές τις αλυσίδες αξιών, είτε παγκόσμιες είτε ευρωπαϊκές, να υπάρχει αποτελεσματική δημιουργία αξίας, αλλά αυτό που μετράει είναι και πόση αξία μπορούμε να ε, έχουμε εμείς ε, από αυτές τις αλυσίδες. Ποιες χώρες και ποιες επιχειρήσεις θα μπορέσουν λοιπόν να εκμεταλλευτούν αυτή την αξία και όπως είπα προηγουμένως, αυτό μπορεί να γίνει μόνο εάν υπάρχουν μοναδικές δυνατότητες ε, βιώσιμες εντός της αλυσίδας αξιών που μας επιτρέπουν να αποκομίσουμε εμείς αξία από όλο αυτό. Και φυσικά αυτό ε, σημαίνει ότι χρειαζόμαστε και δυνατότητες καινοτομίες γιατί αυτή είναι πηγή ε, βιώσιμους μοναδικών δεξιοτήτων που δημιουργούν όχι μόνο αξία αλλά αποκομίζεται και αξία που σημαίνει ότι ο στόχος πολιτικής ε, θα πρέπει να έχει μια αλυσίδα αξία η οποία λειτουργεί πολύ καλά, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και μια ισχυρή βιομηχανική πολιτική που επιτρέπει δυνατότητες καινοτομίας ε, για να μπορέσουμε να αποκομίσουμε αξία από αυτές τις αλυσίδες. Η εμπορική πολιτική λοιπόν πρέπει να συνδεθεί στενά με τη βιομηχανική πολιτική. Αυτό σημαίνει ότι συνολικά ο στόχος της πολιτικής θα πρέπει να είναι η Ευρώπη ε, να είναι ε, τομέας ο οποίος αποτελεί βέλεαρ για να αναπτυχθούν αυτές οι δυνατότητες, να υπάρχει ένα πλαίσιο για να αναπτυχθούν όλα αυτά και βεβαίως θα πρέπει να γνωρίζουμε πού μπορεί να προκύψουν αυτά τα πράγματα που θα είναι πολύ δύσκολο, πού μπορούμε να έχουμε καινοτομία ή πού μπορούμε να έχουμε αποτελεσματικέ πολιτικέ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια οριζόντια πολιτική σε αυτή την περίπτωση. Και τέλο. Είπαμε ότι θέλουμε συνδυασμό εμπορικής πολιτικής και εκτό. Ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν αφορά μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκτό, ε, μετά το Brexit θα είναι πολυμερή τα πράγματα, πρέπει λοιπόν να είμαστε αρκετά ανοιχτοί με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά η ενδοκοινοτική πολιτική σε βιομηχανικό επίπεδο θα πρέπει να επιτρέπει καινοτομία, όπως είπα ήδη αυτή είναι οριζόντια πολιτική αλλά πρέπει να παρακολουθούμε ε, σημαντικούς τομείς ε, για ανάπτυξη που βασίζεται στην καινοτομία, όπου η Ευρώπη πραγματικά έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει βιώσιμες καινοτόμες θέσεις για να αποκομίσει αξία, σίγουρα ο ψηφιακός τομέας, γιατί η ψηφιακή καινοτομία είναι πάρα πολύ σημαντικός μοχλός ε, ανάπτυξης βάσει καινοτομίας, αλλά επειδή είναι και τα ισχυρά χαρτιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, ε, βιοφαρμακευτικός τομέας ε, θα αποτελέσει πολύ σημαντικό μοχλό καινοτομίας ε, στην αλυσίδα αξιών μεταφορές, σίγουρα τα αυτοκίνητα είναι πολύ σημαντικά, αλλά και ο χώρος, ε, ο εναέριος και του διαστήματος, που θα τα συζητήσουμε και αυτά εδώ. Αυτό λοιπόν που έχει σημασία για την βιομηχανική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να έχει ένα ευρωπαϊκό θεματολόγιο πολιτικής και να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε όλους τους τομείς οι οποίοι θα αποτελέσουν και πολύ σημαντικό μοχλό να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό εφαρμίζονται όλες οι συνθήκες ε, πλαίσιο ε, για να αναπτύξουμε αυτούς τους τομείς και αν χρειάζονται συγκεκριμένε παρεμβάσεις πολιτικής για να αντιμετωπίσουμε τους πιθανούς φραγμούς. Αυτά με δύο λόγια, πολύ σύντομα, για τις προκλήσεις που έχουμε στη βιομηχανική πολιτική και τώρα θα πάρουν το λόγο συνάδελφοι. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάντος τώρα, Διευθυντή Διεθνών Σχέσεων στην Business Europe, πρόεδρος της Task Force για το Brexit στην Business Europe. Τώρα είναι μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων για τις διαπραγματεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ινωμένου Βασιλείου. Είμαι ειδική στα μετά εμπορίου, είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ για να μιλήσω για το Brexit. Να σα πω δύο λόγια για τη θέση της Business Europe ποιες είναι οι απόψεις μας ε, γενικά και μετά θα επισέλθω σε κάποια τομεακά και διατομεακά ζητήματα που μπορεί να επηρεάσουν τομείς της οικονομίας, της υπηρεσία, τη βιομηχανία. Άρα, ούτως ή άλλως για μας αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Και τέλος, θα κλείσω μια σύνοψη για να σα πω τι έχουμε κάνει για το Brexit και τι ε, δημοσίευσεις έχουμε πραγματοποιήσει. Όλοι γνωρίζετε ότι ζούμε σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Είδατε τι έγινε στο Σάλτσμπουργκ μετά την, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γνωρίζετε επίσης ότι είμαστε σε μια δραματική καμπή για τον Brexit, για μας, για τις επιχειρήσεις. Το θέμα είναι ότι είμαστε σε μια μετάβαση, θέλουμε μια μετάβαση, δηλαδή έως ότου επιτευχθεί η συμφωνία και προκύψει το νέο πλαίσιο σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου απαιτείται μια σταδιακή μετάβαση από την κατάσταση στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μέλος ως αυτήν στην οποία το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι τρίτη χώρα. Ξεκινάμε λοιπόν από ένα σενάριο στο οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο ξεκινάει από τη σημερινή θέση. Χρειαζόμαστε όμω και μια συμφωνία αποχώρησης. Χωρίς την συμφωνία αποχώρησης δεν θα δρομολογηθεί η μετάβαση μετάβαση και αυτό που προσπαθούν να κάνουν και οι δύο πλευρές. Για μας λοιπόν, έχει σημασία στην παρουσία συγκυρία και επειδή ο χρόνος κυλάει γρήγορα, πρέπει τέλειο Οκτωβρίου, άντε μέσα Νοεμβρίου, να έχουμε εξεύρει λύση όσον αφορά την απόσυρση και να έχουμε λύσει και το θέμα της Ιρλανδίας. Και αυτό για τις επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντικό, αλλιώς δεν έχουμε πλέον και μετάβαση μεταβατική περίοδο, αν θέλετε. Θα ήθελα επίσης να πω συναφώς ότι ενώ ψημελωτικών εξελίξεων, του γίνει δηλαδή τρίτη χώρα του ΕΒ, θα δούμε ποια θα είναι αυτή η κατάσταση, αλλά ε, έχει μεγάλη σημασία οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει να είναι σε στενή σχέση με το ΕΒ και τι επιχειρήσει του. Όμω, και αυτό είναι μια προειδοποίηση που θέλω να απευθύνω, μια πολύ σοβαρή προειδοποίηση, χωρίς, χωρίς σε κάθε περίπτωση να απειληθεί το ενιαίο της εσωτερικής αγοράς. Και αυτό σημαίνει ότι αν το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί βελτιωμένη πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά μετά το Brexit, αυτό θα πρέπει να γίνει με την συνειδητοποίηση από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα έχει λιγότερο έλεγχο στην εσωτερική του αγορά. Το Ηνωμένο Βασίλειο είπε ότι ναι, δεν θέλω να μείνω στην εσωτερική αγορά. Θέλουμε ίσω μια τελωνιακή ένωση. Αυτό είναι δική του επιλογή. Επιλογή τη Βρετανική κυβέρνηση. Όμω δεν θα μπορούν να έχουν φυσικά την ίδια πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά, ίδια με αυτήν που έχουν σήμερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε εδώ σήμερα, διότι οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει θέλουν να προστατεύσουν, να διαφυλάξουν και να προστατεύσουν την εσωτερική αγορά. Την ενιαία εσωτερική αγορά. Ποια λοιπόν τα ζητήματα που έχουμε μπροστά μας. Τέσσερα θέματα θέλω να θέσω, τα οποία επηρεάζουν διάφορε τομείς της βιομηχανίας. Το πρώτο είναι τα τελωνιακά ζητήματα. Όπως γνωρίζετε, προ το παρόν και αυτό είναι η βάση τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ένα ενιαίο εξωτερικό δασμολόγιο. Με άλλα λόγια έχουμε κοινά σύνορα, κοινού δασμούς. Εφαρμόζουμε κοινού κανόνε, τι εμπορικέ σχέσει με, τους, ε, με τις χώρες. Έχουμε ένα ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο. Αυτά είναι η εσωτερική αγορά. Κοινοί κανόνε μεταξύ άλλων. Ήδη κοινωνικά πρότυπα, περιβαλλοντικά πρότυπα, είδου κανόνε για τον ανταγωνισμό, εθνικές πολιτικές κλπ. Αυτό σημαίνει ότι ένα προϊόν που μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα δοκιμαστεί και θα αναλυθεί μία φορά, όπως άλλωστε ισχύει και τα προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν βγει το Ηνωμένο Βασίλειο, όλα αυτά τίθενται ένα αμφιβόλο. Δηλαδή, δεν ξέρουμε τι θα συμβεί με τους δασμούς στο μέλλον. Εάν επιτευχθεί ζώνη ελευθερού εμπορίου θα έχουμε μηδενικούς δασμούς αφωτέρωθων, αλλά δεν υπάρχει ακόμη βεβαιότητα γι' αυτό. Ας πούμε για τα άστρα, μην ξεχνάτε ότι έχουμε υψηλούς δασμούς, 40% αλλά και για βιομηχανικά προϊόντα, για παράδειγμα για τα εφαντουργικά έχουμε 12% για τις τρίτες χώρες, έχουμε 10% για τα οχήματα, διαφόρων τύπων. Οι Αμερικανοί έχουν χαμηλότερου δασμού. Αν λοιπόν πετύχουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και συμφωνήσουμε στου δασμού, τότε οι εταιρείε μα που εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο θα πλήττουν από και ανιστρόφως βεβαίω. Όπω προείπα, θεωρώ ότι θα έχουμε το ίδιο κανονιστικό πλαίσιο στην, Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό σημαίνει ότι αν οι επιχειρήσει θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν του ίδιου κανόνε. Ένα προϊόν θα αρκεί να δοκιμαστεί, να αναλυθεί σε μία από τι δύο πλευρέ. Με την ίδια λοιπόν σήμανση, με την ίδια ετικέτα, ένα προϊόν θα μπορεί να κυκλοφορεί παντού. Εκτό αν βεβαίω δεν καταλήξουμε σε τέτοια συμφωνία ελευθερών μπορεί με τον Ε. το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε προϊόν να αναλύεται, να υποβάλλεται σε δοκιμέ και στι δύο πλευρέ. Και οι επιχειρήσει λοιπόν θα πρέπει πλέον να φροντίσουν να συμμορφώνονται με διαφορετικού κανόνε στι δύο πλευρέ, άρα πλέον επιβάρυνση, φόρτο εργασία, ε, τελειωνιακέ διαδικασίε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, Όμω πέραν όλων αυτών θα έχουμε απλά ελέγχου στα σύνορα. Ξέρετε ότι για παράδειγμα έχουμε υγειονομικά και φυτογειονομικά μέτρα πολύ αυστηρά για κάθε προϊόν που εισάγεται από τρίτη χώρα. Κάθε προϊόν το οποίο εισάγεται από τρίτη χώρα πρέπει να ελέγχεται για να διασφαλίσουμε ότι συνάδει, συμμορφώνεται με τους ενωσιακούς κανόνες, συν όλη η γραφειοκρατία κλπ. κλπ. Άρα, εάν δεν επιτευχθεί η συμφωνία με τον Ηνωμένο Βασίλειο, είναι βέβαιο όπως είπε και η προλαλήσασα, θα υπάρχουν θα υπάρξουν πολύ σημαντικές επιπτώσεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες μεταξύ των δύο πλευρών, διάφορα προϊόντα για να μπουν και να βγουν θα αντιμετωπίζουν αυτά τα εμπόδια, θα έχουμε τελωνικούς ελέγχους, επιπλέον δοκιμές, επιπλέον αναλύσει και όλα αυτά αυξάνουν το κόστος. Αλλά όχι μόνο αυτό. Θα αυξηθεί και ο ρυθμός των διαδικασιών που θα πετούνται στα σύνορα. Κανόνες προέλευσης. Κανόνες καταγωγής, μάλλον. Ε, ξέρω ότι δεν αρέσει πολλούς, αλλά είναι προϋπόθεση για την απαλλαγή από δασμούς. Με άλλα λόγια, πρέπει επαρκές παραχθέν περιεχόμενο, ποσοστό περιεχομένου να έχει παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απαλλαγή, α πούμε, για τα αυτοκίνητα. 55% της προστιθέμενης αξίας πρέπει να έχει παραχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να χορηγηθεί προτιμησιακή μεταχείριση και αντίθέτω. για να μην επιβληθεί δηλαδή δασμός. Και αυτό είναι πρόβλημα διότι σήμερα τα αυτοκίνητα φτιάχνονται με συνεισφορές υλικών από πολλές διαφορετικές χώρες. Τα πάρτια τα οποία θα προέρχονται τα αυτοκίνητα τα οποία θα περιέχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να συμμορφώνονται με αυτόν τον κανόνα. Πράγμα το οποίο, το οποίο σημαίνει με τη σειρά του ότι οι εφοδιαστικέ αλυσίδε θα αλλάξουν στην περίπτωση που δεν συμμορφώνονται με την απέτηση αυτή, για να μπορούν δηλαδή να απαλλαγούν τα αυτοκίνητα από το δασμό. Να θυμίσω κάτι πολύ σημαντικό. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συμφωνήσει με Κορέα, με Καναδά, και χρησιμοποιούμε υλικά από αυτές τις χώρες. Αν αύριο το Ηνωμένο Βασίλειο θεσπίσει διαφορετικούς κανόνες, εάν δεν υιοθετήσει το Ηνωμένο Βασίλειο, δηλαδή 100% τους κανόνες τους ευρωπαϊκούς, τότε θα επηρεαστούν τα ενδιάμεσα προϊόντα, τα απάρτια και ανταλλακτικά τα οποία εισάγονται από το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό θα επηρεάσει, όπως ξαναείπα, την εφοδιαστική αλυσίδα. Κανονιστικό πλαίσιο. Κάποιοι κανόνες, κάποιοι τομείς, με συγχωρείτε, λιγότερο περισσότερο θα επηρεαστούν. Εδώ μιλούμε για περιβαλλοντικά πρότυπα, κοινωνικά πρότυπα και θέλουμε να ισχύσουν ήδη κανόνες για όλους, όχι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Για να υπάρχει και διαφανής ισότιμος ανταγωνισμός. Η ροή των δεδομένων. Και εδώ θα επηρεαστούν διάφοροι τομείς γνωρίζετε τον κανονισμό GDPR περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει προφανώς, συμμερίζεται τους ίδιους κανόνες, αλλά από τη στιγμή που θα γίνει τρίτη χώρα, όπως φαντάζεστε, με βάση τους ενωσιακούς κανόνες, το Ηνωμένο Βασίλειο πλέον δεν θα συμμορφώνεται. Θα χρειαστεί λοιπόν περί επάρκειας απόφαση adequacy decision ή ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διπλωδρών. Αυτό μπορεί να πάρει χρόνο, θα πάρει χρόνο δηλαδή μέχρι να εξασφαλίσουμε αυτή την απόφαση. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι εντωμεταξύ θα κυριαρχεί μεγάλη βεβαιότητα για του συναλλασσομένου. Έρευνα και ανάπτυξη, να μην τα ξαναπούμε. Έχετε ένα εργαστήριο αφιερωμένο σε αυτό, αλλά σίγουρα είναι ένα τομέα ε, στον οποίο θα θέλαμε να διατηρήσουμε στενέ σχέσει με το Ηνωμένο Βασίλειο. Εδώ βλέπετε δύο δημοσιεύσει για το Brexit διατρέχει που έχουμε δημοσιεύσει για να προετοιμάσουμε τις επιχειρήσεις που θέλουμε να είναι έτοιμες. Δεν ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω πού πηγαίνουμε, δεν ξέρω ποια θα είναι η μελλοντική σχέση Ευρωπαϊκή Ένωση Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο δυνατό σενάριο. Πρέπει οι επιχειρήσει να είναι ενημερωμένε για το τι μπορεί να συμβεί και αυτό είναι και το πιο δύσκολο, ειδικά για τι μικρομεσαίε. Μέρο ένα μάλλον από τους στόχους της Business Europe είναι να προετοιμάσει τις επιχειρήσεις ενημερώνοντας για τους τομείς στου οποίους ε, πιθανότερα θα δούμε τι επιπτώσει από τον Brexit. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά κυρία Σάντο. Ο επόμενος ε, τώρα ο μιλητή είναι ο κύριο Τορτορά, ο οποίο από τον Ιούνιο του 2016 έχει αναλάβει ω διευθυντή του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Πολιτική του Διαστήματο ε, και από ό,τι γνωρίζω προηγουμένω ε, ήταν ο επικεφαλή τη Οποσπονδία τη Ευρωπαϊκή Βιομηχανία Διαστήματο, ε, ενώ από το 2004 έως το 2007 ήταν επικεφαλή του γραφείου τη Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία στην Βόρεια Αμερική και επίση ακόλουθο στην πρεσβεία τη Γαλλία για τα ζητήματα διαστήματο και αεροναυπηγική στη Ουάσιγκτον. Έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ και με, χαρά μου παρευρίσκομαι σήμερα εδώ για να σα ε, αναφερθώ στην πολιτική διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καταρχήν να σα πω δύο λόγια σε ό,τι αφορά το Ινστιτούτο μα, το οποίο έχει την έδρα του στη Βιέννη και είναι πραγματικά ε, μοναδικό σε ευρωπαϊκό think tank, το οποίο πραγματικά είναι αφιερωμένο 100% στα ζητήματα διαστημικής ε, πολιτική και στις σχετικέ. Ε, σκέψεις που θα πρέπει να κάνουμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο και το διάστημα. Επιτρέψτε μου να κάνω καταρχήν κάποια, μια γενική περιγραφή, αν θέλετε, του ε, ποια είναι τα ειδικά χαρακτηριστικά τη ε, παρουσία του Ενωμένου Βασιλείου σε αυτό το τομέα. Καταρχήν, να σα υπενθυμίσω ότι ε, το Ενωμένο Βασιλείο συμμετέχει σε μια σειρά από διακυβερνητικέ οργανώσει όπω ο ε, Ευρωπαϊκό Οργανισμό του Διαστήματο, η Ευρωπαϊκή Οργάνωση για την Μετάλλευση Μετρολογικών Δορυφόρων, η UMETSAT και ούτω καθεξή. Και αυτό θα συνεχίσει και μετά τον Brexit. Ωστόσο, θα ήθελα επίση να σα τονίσω ότι το ΕΒ. Βασίλειο ανέκαθεν παραδοσιακά εστιάζει και στις επιχειρήσεις και στις εφαρμογές, τα application ε, και μάλιστα περισσότερο μάλλον από οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος ε, τη σήμερον ημέρα. Και αυτό σημαίνει ότι συμμετέχει σε περιορισμένο βαθμό στο Αριάνε και στις επαντρωμένες ε, διαστημικές πτήσεις καθώς κάτι τέτοιο δεν ευθυγραμμίζεται με το στρατηγικό όραμα του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς το πώς δηλαδή θα πρέπει να δραστηριοποιείται η βιομηχανία διαστημική του σε αυτό το τομέα. Επίσης θα ήθελα να σας τονίσω ότι ε, το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε, είναι πολύ ευαίσθητο σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, δηλαδή εδώ συμμετέχει πολύ ενεργά στις, στις σκέψεις και στη χάραξη πολιτικής σε αυτό το τομέα και αν αναλογιστούμε δηλαδή αυτή την προοπτική της εξόδου της, το κύκλο των κρατών μελών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, στο μέλλον, τότε θα οδηγηθούμε στο συμπέρασμα ότι θα υπάρξει κάποιο αντίκτυπο. Και επίση, κάτι ακόμα που θα ήθελα να αναφέρω είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι, έχει την πιο φιλελεύθερη προσέγγιση σε ό,τι αφορά το διάστημα σε σύγκριση με όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και αν κάποιο δεν με πιστεύει σε σχέση με αυτό το τελευταίο σημείο, σα δείχνω εδώ ένα διάγραμμα το οποίο περιλαμβάνεται σε μια έκθεση την οποία θα δημοσιεύσουμε μέσα στις επόμενες εβδομάδες και βλέπετε λοιπόν εδώ σε αυτό το διάγραμμα ποια είναι η κατανομή ε, των ιδιωτικών επενδύσεων στον τομέα του διαστήματος. Και ειδικότερα δε επενδύσει στο πλαίσιο αυτού του επωνομαζόμενου New Space. Εδώ βλέπετε λοιπόν ότι με μεγάλη διαφορά από τους υπολείπους ε, στο, το Ηνωμένο Βασίλειο είναι εκείνο στο οποίο λαμβάνουν η χώρα η πλειοψηφία όλων αυτών των δραστηριοτήτων, των επενδύσεων δηλαδή, το 1 τρίτο δηλαδή το συνόλου των σχετικών δράσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό δηλαδή μας λέει πολλά ως προς ε, ε, το ποια είναι η ιδιαιτερότητα του Ηνωμένου Βασιλείου ως μέλος σε αυτές τις δραστηριότητες και θα σας αναλύσω και τις δικές μου σκέψεις σε σχέση με αυτό, αλλά και το ποιος θα μπορούσε να είναι ο πιθανός αντίκτυπος της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από ε, την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια από τα διάφορα σημαντικά προγράμματα του διαστήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ξεκινάω με το Κοπέρνικους. Εδώ σας ε, υπενθυμίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πολύ ε, πιθανόν θα συνεχίσει την συμμετοχή του στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό του Διαστήματος, του EUMETSAT, στο ε, Κέντρο Μεσοπρόθεσων Μετρολογικών Προβλέψεων, το Mercator ε, και ούτω καθεξής. Και αυτό σημαίνει ότι θα έχει πρόσβαση σε ένα μεγάλο όγκο δεδομένων. Αλλά και το Κοπέρνικους βασίζεται ε, σε μια φιλοσοφία ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι θα υπάρχει ροή δεδομένων. Εντάξει, φυσικά μπορούν να υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί σε ό,τι αφορά τα, ε, τους χορηγούς και ίσως να υπάρξουν κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την ευρυζωνική πρόσβαση στα σχετικά δεδομένα, αλλά ε, εκείνο που είναι το βασικό ζήτημα, είναι η δυνατότητα της Βρετανικής βιομηχανίας να, να, να, συνεχίσει να συμμετέχει στο πρόγραμμα Κοπέρνικους και στο μέλλον. Και ε, όταν εδώ έχουμε τα σχετικά σύμβολα που συνάπτονται από την πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και όταν έχουμε την εφαρμογή των κανόνων των δημοσίων συμβάσεων τη ε, προμήθεια δηλαδή, τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εκεί θα υπάρξει αυτή η ιδιαιτερότητα και εδώ αναφέρομαι σε ό,τι αφορά το Κοπέρνικο. Αλλά ο Κοπέρνικο έχει μια ιδιαίτερο, ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα συνεργατικό, οπότε νομίζω πω θα είναι προ το συμφέρον όλων των συμμετεχόντων να συνεργαστούν και να συνεχίσουν να εργάζονται ε, σε μία βάση όσο το δυνατόν ευρύτερη ε, συμμετοχή. Γιατί όσο μεγαλύτερη είναι η βάση των συμμετεχόντων, ο αριθμό των συμμετεχόντων, ε, τόσο μεγαλύτερο το όφελο για το πρόγραμμα. Άρα λοιπόν αναμένω πω θα συναυτούν κάποιε συμφωνίε έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αρμονική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτό το πρόγραμμα και στο μέλλον. Αλλά βέβαια αυτή είναι δική μου εκτίμηση, δική μου πρόβλεψη. Τώρα έρχομαι στο ε, τομέα της ε, ασφάλειας, της διαστημικής ασφάλειας. Ε, το ζήτημα που τίθεται εδώ είναι η δυνατότητα ε, συμμετοχής του Βασιλού στα σχετικά προγράμματα SST και SSA σε ό,τι αφορά την παρακολούθηση και τον έλεγχο αλλά και την καταστασιακή γνώση των καταστάσεων από την πλευρά των συμμετοχών. Ε, υπάρχουν λοιπόν κάποια πρακτικά ζητήματα, αλλά δεν βλέπω ε, πως ε, να υπάρχει ιδιαίτερο λόγο για ανησυχία, γιατί θα υπάρξουν περιθώρια και μεσοπρόθεσμα σε ό,τι αφορά διαπραγμάτευση, αλλά και επειδή δεν υπάρχουν πολύ σημαντικά περιουσιακά στοιχεία του Ηνωμένου Βασιλείου σε αυτά τα προγράμματα. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με τη Γερμανία και τη Γαλλία, οι οποίε έχουν επενδύσει σε μεγάλο βαθμό στο σύνοδο δηλαδή, σε σύγκριση με το σύνοδο των 27 κρατών μελών σε αυτά τα προγράμματα. Από εκεί και μετά έχουμε ε, την Νάσαντ ε, και εδώ αναφέρομαι δηλαδή γενικότερα σε αυτήν και σε άλλους ε, μεγάλους παίκτες, ας το πούμε έτσι, της βιομηχανίας της διαστημικής του Ηνωμένου Βασιλείου, οι οποίοι στο πλαίσιο ενός συνεργατικού πλαισίου ανταλλάσσουν μεταξύ τους πληροφορίες σε ό,τι αφορά τις γεωστατικές τροχές, για τους στόχους δηλαδή της αποφυγής συγκρούσεων και ούτω καθεξής. Όλα αυτά λοιπόν δεν νομίζουμε πως θα ποστούν κάποια αρνητική συνέπεια από τον Brexit. Και τέλος, σε αυτόν τον τομέα υπάρχουν ε, ορισμένες υπηρεσίες οι οποίες διατίθεται από, το, ε, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικότερα από το ε, Υπουργείο Άμυνας, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι εν λόγω υπηρεσίες θα συνεχίσουν να παρέχονται σε εμπορική βάση και ε, μακροπρόθεσμα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Άρα λοιπόν, σε σχέση με αυτό το ζήτημα, δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερη ανησυχία. Τώρα, περνάω στις ε, κυβερνητικέ δορυφορικέ επικοινωνίε, τα GovSatcoms. Ε, εδώ μιλάμε για ένα από τα νέα προγράμματα τα οποία έχουν προταθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, αυτό ο τομέα των κυβερνητικών δορυφορικών επικοινωνιών, δηλαδή για τι ασφαλείς δορυφορικέ επικοινωνίες, είναι ο μοναδικός τομέας στον οποίο στον, οποίο έχει πράγματι το Ηνωμένο Βασίλειο εφαρμόσει μια εθνική διαστημική πολιτική. Δηλαδή, επί σειρά ετών έχουν πράγματι ε, μέσω τη σειρά Skynet που βρισκόμαστε τώρα στη Skynet 5 και ετοιμάζεται το Skynet 6, μια σειρά λοιπόν από ε, τέτοιου είδου ε, ε, υπηρεσίε, δράσει δηλαδή κυβερνητικών επικοινωνιών και ε, γενικότερα σε αυτό το πλαίσιο να πούμε ότι η βιομηχανία ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, συμμετέχει και στα, μάλλον θα συνεχίσει, δεν ανησυχούμε ότι θα συνεχίσει να συμμετέχει, συμμετέχει στις επιχειρηματικές δραστηριότητες των GeoSatcoms και για αυτούς λοιπόν τους λόγους το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν μας δημιουργεί ιδιαίτερες ανησυχίες. Και έρχομαι τώρα στο Γαλιλαίο. Ε, και εδώ να σας υπενθυμίσω ότι αρχικά το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ταχθεί εμφαντικά κατά αυτού του προγράμματος και όταν τελικά αποφασίστηκε ότι θα τρέξει ε, κατάφεραν να τοποθετήσουν ε, στον πυρήνα αυτού του προγράμματος στη δική τους βιομηχανία. Στον πυρήνα δηλαδή του PRS, του Public Regulated Service. Και εδώ πρόκειται για το πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί τη μεγαλύτερη, αν θέλετε, σύγχυση ή ε, τις μεγαλύτερου μεγαλύτερους φόβους σε ό,τι αφορά τη μελλοντική συμμετοχή του ΕΒ. Βασιλείου. Το βασικό συμπέρασμα λοιπόν που θα μπορούσαμε να αντλήσουμε από αυτή την κατάσταση είναι το ότι αν θέλουμε να καταδείξουμε το ε, ποια είναι η συνάφεια του ΕΒ Βασιλείου για το Γαλιλαίο, ε, νομίζω πως αν ρίξουμε μια ματιά σε όλες τις σχετικές συζητήσεις που γίνονται θα διαπιστώσουμε ότι όλες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι πραγματικά έχει μεγάλη αξία αυτή η συμμετοχή. Όλα τώρα τα ε, μη στρατιωτικά σήματα, δηλαδή συμπεριλαμβανομένου και του έγκνους, θα συνεχίσουν να είναι διαθέσιμα και στο ένωμα Βασίλειο. Ε, αλλά από εκεί και μετά η πρόσβαση στο Public Regulatory Service, στο PRS, ε, παραμένει σε κρεμότητα. Δεν γνωρίζουμε δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί και επίση εκείνο που ανησυχεί είναι η μελλοντική ε, συμμετοχή της ε, Διαστημική μηχανής του Ηνωμένου Βασιλείου στις μελλοντικές εξελίξεις. Εδώ καταρχήν ε, τίθεται το ερώτημα της πρόσβασης στο ΣΥΝΟ και νομίζω πω εδώ το σχετικό ερώτημα είναι εύκολο να απαντηθεί, αλλά το δεύτερο ερώτημα και το πιο δύσκολο είναι η συμμετοχή της ε, Βρετανικής βιομηχανίας στον πυρήνα, αν θέλετε, της διαχείρισης του συστήματος. Δηλαδή, θα πρέπει να χορηγηθεί σε αυτή τη βιομηχανία, τη Βρετανική και στο μέλλον, ε, ένας τέτοιος ρόλος, ε, συμμετοχής δηλαδή στον πυρήνα της διαχείρισης ή όχι. Και κλείνω εδώ δώντας κάποια συμπεράσματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν αυτήν την υπόθεση, θέλετε, το, το γενικότερο πρόβλημα της συμμετοχής στη διαστημική πολιτική του της, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου ε, μετά το Brexit. Να πούμε ότι ε, το όλο ζήτημα δεν αντιστοιχεί ε, στη, στον, στο πραγματικό μέγεθος αυτού του κλάδου. Ε, δηλαδή, από οικονομική άποψη δεν τίθεται ιδιαίτερο ζήτημα, αλλά βέβαια το δεν είναι αμυγός οικονομικής φύσης ε, το πρόβλημα. Από εκεί και μετά βλέπουμε πως ε, έχει αναλάβει εδώ ηγετικό ρόλο το Ηνωμένο Βασίλειο σε ό,τι αφορά την, ε, βιομηχανία, την διαστημική βιομηχανία και παρόλα αυτά κατάφερε να αναλάβει το 17% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων στον Καλιλαίο και επίσης η βιομηχανία του Ηνωμένου Βασιλείου είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένη προς τις εξαγωγές. Οπότε υπάρχει ένας κίνδυνος εκεί. Και παρότι λοιπόν Ευρωπαϊκός Οργανισμός Οργανισμό και έρευνα και τεχνολογία δεν θα υποστούν αρτικε συνέπειε από το Brexit. Ε, το ζητούμενο είναι το κατά πόσο κάτι τέτοιο θα είναι ικανό να διατηρήσει την κρίσιμη μάζα της βιομηχανίας ε, στο Ενωμένο Βασίλειο. Δηλαδή, ειδικότερα στο πλαίσιο της συμμετοχής ε, στο ISS, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, όπου ουσιαστικά άπαξα πάνω χώρα τα προγράμματα. Και αυτή είναι γενικότερα και η πρακτική που ακολουθείται και στα διάφορα προγράμματα ε, όπως το Γαλιλαίο και το Κοπέρνικους. Από εκεί και μετά ίσως να αντιμετωπίσει το ΕΒ ορισμένα προβλήματα σε ό,τι αφορά τις εφοδιαστικές αλυσίδες, δηλαδή την πρόσβαση σε κρίσιμες ε, τεχνολογίες, αλλά και πρόσβαση σε ό,τι αφορά το ταλέντο, το αντίστοιχο δηλαδή ε, ανθρώπινο δυναμικό. Και τέλος, ε, ε, σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ασφάλειας και άμυνας, θα πρέπει αυτά να αντιμετωπιστούν με έναν συνεκτικό τρόπο με βάση τα όσα ευρύτερα θα συμφωνηθούν στο επίπεδο συνεργασίας σε ζητήματα ασφάλειας και άμυνας με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, όπως σας είπα ήδη, η Βρετανική πλευρά συνέβαλε στη διαμόρφωση της πολιτικής στο διάστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ασφάλεια και άμυνα και πιθανότατα το διάστημα θα αποτελέσει μια πρώτη, πρώτη ένδειξη, αν θέλετε, για τον ε, τρόπο συνεργασίας ε, που θα βρουν μεταξύ τους ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Θα ξεκινήσει τώρα η διαδικασία ερωτήσεων και απαντήσεων από τα μέλη και η πρώτη είναι η κυρία Βαμπρέντα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο. Ζήτησα το λόγο ε, όχι για να μιλήσω εξ ονόματός μου, θα μιλήσω εξ ονόματος του καλή συναδέλφου Τερέζα Γκρίφιν. Θέλω να διαβάσω μία δήλωση και μία ερώτηση. Δεν μπορεί να είναι εδώ, έχει μια διάσκεψη στην πρωτεύουσά της. Ε, θα μιλήσω λοιπόν εξ ονόματος της Τερέζα Γκρίφιν που ε, είναι ε, αρμόδια για τα θέματα αυτά από τους εργατικούς. Το Brexit ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί αλλά ε, νιώθουμε τον αντίκτυπο. Σύμφωνα με την έκθεση για IPPR για την Βόρεια Αγγλία, ο Βορράς θα επηρεαστεί περισσότερο από τον Νότο βλέπουμε απόλυση της τάξη του 2,5% του ΑΕΠ στην βορειοδυτική οικονομία, εάν επιλέξει ε, μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου. Αν έχουμε μια μορφή ε, συμφωνία σαν τον Καναδά θα έχουμε 3,5% και το ποσοστό είναι πολύ μεγαλύτερο αν έχουμε ε, σκληρό Brexit, δηλαδή δεν υπάρξει συμφωνία. Το, το οποίο λοιπόν είναι καταστροφικό και η ενιαία αγορά ε, έχει 3 εκατομμύρια θέσει εργασία που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 1,5 δισεκατομμύριο κύκλο εργασιών και πολύ μεγάλο ποσοστό εργαζομένων προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι εργαζόμενοι χάνουν ήδη τις θέσει εργασία τη λόγω των μειώσεων προσωπικού ή της ε, μετεγκατάσταση λόγω του Brexit. Το είδαμε αυτό στι αυτοκινητοβιομηχανίε. η Jaguar, η Land Rover ανακοίνωσαν προσφάτω ότι λόγω της, ε, των συνεπειών του Brexit θα περικόψουν την παραγωγή και αν υπάρξει Brexit χωρί συμφωνία, μπορεί όλη η παραγωγή να πρέπει να μεταφορθεί στη Σλοβακία και πιθανόν να χαθούν 14.000 θέσει εργασία και 250.000 θέσει εργασία στην αλυσίδα ε, προμηθειών. Το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα σχετικά προγράμματα και αν υπάρξει αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου φυσικά θα μπορεί να επηρεάσει πολύ λιγότερο ε, τα διαστημικά προγράμματα, λιγότερη πρόσβαση σε δορυφόρους, σε διαστημική τεχνολογία κλπ. Ε, και ε, υπάρχει πρόβλεψη για συρρήκνωση κατά 1,8%. Η Airbus είπε ότι θα μεταφέρει συμβάσεις για τους δορυφόρους και τα συστήματά τους από το Ηνωμένο Βασίλειο σε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συμφωνία λοιπόν ε, χωρίς ε, μάλλον, εάν δεν υπάρχει συμφωνία και έχουμε αποχώρηση απλώς, ε, τότε θα υπάρχει ε, πανεξέταση της πολιτικής τους και χάνονται θέσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, οι μισές εξ αυτών στην Ουαλία και έχουμε και πάνω από 100.000 θέσεις εργασίας στην αλυσίδα προμηθειών. Η κυρία Γκρίφιν, λοιπόν, κάνει μια έκκληση την οποία κατανοώ απολύτως πώς μπορεί να το εξηγήσει αυτό ε, στην περιφέρειά της, ε, όταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι κινδυνεύουν να χάσουν τις θέσεις εργασίας τους και ε, μειώνεται η παραγωγή. Και αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Βανμπρέμπτ. Θα ακούσουμε κάποιες ερωτήσεις και μετά το πάνελ θα έχει δυνατότητα να απαντήσει. Ο κύριος Τένικα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τις απόψεις που εκφράστηκαν από τους ομιλητές μας σήμερα. Και έχω την εξής ερώτηση. Μάλλον η ερώτηση απευθύνεται στη Βρετανική κυβέρνηση και όχι σε εσά. Ξέρουν ποιο θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της περιπέτειας. Έχουν τα σωστά στοιχεία κατά νου. Όσο συγητής για τον ε, ορίζοντα Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με προσέγγισαν ε, Βρετανοί, πανεπιστημιακοί, ερευνητικά ιδρύματα της Βρετανίας, ε, όλοι λίγο πολύ. Το θέμα είναι τι θα γίνει με τη συνεργασία μας. Πού θα βρισκόμαστε και ποια θα, είναι θέση θα έχουμε εμείς ε, στο πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Εγώ πάντα απαντώ, είστε κράτος μέλος. Αν αποφασίσετε να αποχωρήσετε, τότε να είστε βέβαιοι ότι υπάρχουν ε, κατάλληλες προϋποθέσεις και συνθήκες στο λεγόμενο διαζύγιο. Συνάντησα τον κύριο Μπαρνιέ, παρακολούθησα πολύ προσεκτικά αυτό που είχε να πει και ουσία, στην ουσία μας είπε ε, στο 100% αυτά που ε, αναπτύξατε εσείς, ε, γιατί πρόκειται για στοιχεία. Ε, δεν αναφερόμαστε σε διάφορα πιθανά σενάρια για το τι θα συμβεί ε, σε, σαν να ήταν λογοτεχνία επιστημονικής φαντασίας. Για μένα λοιπόν υπάρχει μόνο ένα ερώτημα ουσιαστικά. Λέτε ότι θα πληγεί η Βρετανική βιομηχανία, θα υπάρξει πρόβλημα με τους πολίτες, ε, θα πληγεί το Βρετανικό εμπόριο. Το γνωρίζουν αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, όλοι αυτοί οι εκπρόσωποι οι ε, Βρετανοί πολίτες στην ουσία γνωρίζουν τις συνέπειες, διότι εμείς συζητούμε εδώ στις Βρυξέλλες. Μεταδίδεται και ζωντανά στο διαδίκτυο η συνεδρίαση. Αλλά δεν ξέρουμε πόσοι Βρετανοί μας παρακολουθούν. Ε. Γνωρίζουν ε, λοιπόν ποιες θα είναι οι συνέπειες σε έξι μήνες μετά το Brexit. Τι θα γίνει μετά το πέρας της προθεσμίας. Ευχαριστούμε κύριε Νίκα. Και τέλος ο κύριος και έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω τη μητρική μου. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή την πολύ αναλυτική περιγραφή των διαφόρων θεμάτων και προβλημάτων που μπορεί να ανακύψουν ε, ε, λόγω του Brexit. Πιστεύω ότι το πρόγραμμα Κοπέρνικους μπορεί να διευθετηθεί απλά, όπως μας είπατε, βάσει εμπορικής συμφωνίας. Αλλά η ερώτησή μου αφορά το πρόγραμμα Γαλιλαίο. Δεν ε, θεωρώ ότι υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το PRS. Θα μπορούσε να γίνει επί τη βάση ε, εμπορική συμφωνίας, αλλά τον Γαλιλαίο αυτό καθε αυτό αναπτύχθηκε πάρα πολύ και είναι τμήμα των συστημάτων ασφαλείας και πιστεύω ότι θα ήταν κρίμα το Ηνωμένο Βασίλειο ξαφνικά να θεωρείται τρίτη χώρα, διότι είναι πολύ σημαντική χώρα για αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Η ερώτηση μου είναι Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος έξυπνος, λογικός τρόπος ώστε να προχωρήσουμε και το Ηνωμένο Βασίλειο να μην θεωρείται τρίτη χώρα, αλλά να συμμετέχει ενεργά στον Καλλιλέο, διότι τον Καλλιλέο με τον τρόπο που εφαρμόζεται τώρα ε, αναμένεται να γίνει ένα πάρα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα και εγώ θεωρώ ότι θα αποτελέσει πολύ σοβαρό πρόβλημα ε, να μην μπορέσουμε να επιλύσουμε την κατάσταση για αυτό το πρόγραμμα το οποίο είναι και τόσο δαπανηρό. Βρίσκετε εσεί ότι υπάρχει κάποια λύση. Να ακούσουμε τους ομιλητές για κάποιες πολύ σύντομε παρεμβάσεις και να κλείσουμε. Δυστυχώ πολύ σύντομα, γιατί είναι σημαντικό το θέμα. Όπως και ο Σνίκεν και η Φανμπρέντ. Πολλοί προσπαθούν να υπολογίσουν τι απολύσει του Ηνωμένου Βασίλειου. Ποια θα είναι η ζημία. Και τι θα γίνει με την εμπορική πολιτική. Και τι θα γίνει με την βιομηχανική πολιτική εντός των σύνορων και εκεί υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα. Γιατί μετά εμπόριο και βιομηχανική πολιτική είναι αλληλεύεται τα πράγματα και οι αναπροσαρμογές που θα χρειαστεί να γίνουν αυξάνουν το κόστος. Τώρα για τους 27 και την βιομηχανική πολιτική ε, να πω ότι μην νομίζετε ότι οποιαδήποτε απώλεια για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι κέρδος για μας αναγκαστικά. Έχουν γίνει πολλές μελέτες για τα αρνητικά, για τις αρνητικές επιπτώσεις στον Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και εμείς θα αντιμετωπίσουμε μια βεβαιότητα. Θα εξαρτηθεί όλο αυτό και από το ποια θα είναι η βιομηχανική πολιτική του Ηνωμένου ποια θα είναι η βιομηχανική πολιτική των 27 κλπ. Οπότε, οι 27 πρέπει να πάρουν μια απόφαση τι είδους πολιτική και τι είδους πολιτικές θέλουν μετά το Brexit λόγω του αλληλένδετου των αλυσίδων αξίας. Θέλουμε μια πολιτική ανοιχτή προς τα έξω η οποία θα συνδυάζεται με μια στιβαρή βιομηχανική πολιτική για να διατηρήσουμε μια Ευρώπη που θα είναι Ευρώπη της καινοτομίας. Δυστυχώς τώρα η μία εφοδιαστική αλυσίδα, το ένα πλαίσιο θα γίνει δύο. Εμείς πρέπει να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα παραμείνουμε προσκολλημένοι σε μια ανοιχτή πολιτική και θα συνεχίσουμε να επενδύουμε έτσι περαιτέρω στην βιομηχανική πολιτική η οποία θα αποσκοπεί στην καινοτομία. Το αν ο κόσμος τη Βρετανία γνωρίζει οι επιχειρηματίε γνωρίζουν. Πάντω, ε, μεταξύ των μικρομεσαίων, κάποιοι ξέρουν, κάποιοι δεν ξέρουν, αλλά και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιοι δεν ξέρουν ότι δεν θα μπορούν να εξάγουν προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Οπότε εμεί πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερώνουμε για τι εφοδιαστικέ αλυσίδε. να ξέρουν τι χρειάζεται έτσι ώστε τα προϊόντα να συνεχίσουν να κινούνται, αν και κάποιοι πολλούν στη Γαλλία, στην Γερμανία, χωρίς να ξέρουν ότι τα προϊόντα αυτά ενσωματώνονται σε προϊόν που πήγαινε τελικά στη Βρετανία. Κοιτάξτε, μια εμπορική συμφωνία σε κάθε περίπτωση είναι περιορισμένου εύρου. δηλαδή δεν καλύπτει την καινοτομία, για παράδειγμα, τα έργα καινοτομία. Μην νομίζετε ότι μια απλή εμπορική συμφωνία αποτελεί πανάκια. Το ξέρουμε και εμείς το Ηνωμένο Βασίλειο ότι φυσικά μπορούμε να υπογράψουμε μια εμπορική συμφωνία, αλλά χρειάζονται και πολύ περισσότερα. Δεν είναι μόνο το εμπόριο, με άλλα λόγια. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο θέλει να συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο Horizon, στο Κοπέρνικος κλπ. Πρέπει να το πάρει απόφαση ότι θα πρέπει να τηρήσει τους ίδιους κανόνες, τους ευρωπαϊκούς κανόνες. Αλλιώς θα υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός. Αυτό δεν το θέλουν οι επιχειρήσεις μας. Φυσικά σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενώς με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό θα εξαρτάται από τον Ηνωμένο Βασίλειο και την κυβέρνησή του. Αλλά σε κάθε περίπτωση με την προϋπόθεση του σεβασμού των ευρωπαϊκών κανόνων. Ευχαριστώ κύριε, κύριε Τουρτούρα. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις να το εξή. Με το Brexit, η βασική επιπτώση είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται τρίτη χώρα. Φυσικά θα παραμείνουμε καλοί φίλοι, έτσι. Αυτό έχω πρότεινει άλλωστε. Και από εκεί πέρα υπάρχουν πολλές διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις, συμφωνίες για να διασφαλιστεί η συνέχιση τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στα διαστημικά προγράμματα. Όπω σωστά είπατε όμω, έχουμε τα PRS. Γιατί αυτό σχεδιάστηκε με γνώμονα την κυριαρχία. Φυσικά, όταν έχουμε φίλους ε, του κόλλουμε σπίτι μα, αλλά δεν του δίνουμε τα κλειδιά του σπιτιού μας, για να το πω μεταφορικά. Και αυτό το είδο την πολιτική απόφαση πρέπει να λάβουμε. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία, λέει πρόεδρο. Κλείνουμε λοιπόν με αυτό. Ευχαριστώ τους ομιλητέ, ευχαριστώ που ήρθατε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι εισηγήσει σα. Ευχαριστώ και του βουλευτέ. Γεια σας. Καλησπέρα κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Α περάσουμε λοιπόν στις ψηφοφορίε μας. Να σας παρακαλέσω λοιπόν να βάλετε τις κάρτες ψήφου σα στη σχισμή, στο μηχάνημα και να κάνουμε τη δοκιμαστική ψηφοφορία μας λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία. yet. Maybe could be slightly more. Δεν ξέρω αν είμαστε όλοι εδώ 44, τα δύο τρίτα. Τα δύο τρίτα λοιπόν του αριθμού των μελών. Καλώς. Τι να κάνουμε. Πέρασε στις ψηφοφορίες λοιπόν. Παρακαλώ. Ναι, κύριε Πρόεδρε, σηκώνω το χέρι μου για να μην χρειαστεί να πάω να φέρω την κάρτα μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς λοιπόν. Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2019 με εισηγητή τον ε, κύριο Γιάννη Και μιλάμε εδώ για όλα τα τμήματα, έτσι, από τον οποίο θα ψηφίσουμε. Σημασία τροπολογία υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προσθήκε στην συμβαστική τροπολογία. να υπέρ, κατά, απόχέ, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, ας ελέγξουμε τη 5. Ελέγχουμε λοιπόν την τροπολογία 5 ηλεκτρονικά, πέρας, απορρίπτεται. 6 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Προσθήκη στην συμβαστική 3 υπέρ, συγγνώμη 4 υπέρ, κατά. Ας ελέγξουμε, ας ελέγξουμε. Την προσθήκη λοιπόν συμβαστική τροπολογία 4, ηλεκτρονικά. Πέραση τη φοφορία, Απορρίπτεται. Α, όχι. Εγκρίνεται, εγκρίνεται. «25 περ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 26 περ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 28 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 29 υπέρ, κατά. 29 ξανά. Ας, ας ε, την αλλάξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Η τροπολογία 29. Γιατί δεν είμαι σίγουρος. Πέρα της ηλεκτρονικής προφορίας. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ξεκάθαρο και σας ζητώ συγγνώμη. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην ψηφοφορία λοιπόν, ονομαστική. Α, επί της διαδικασίας, παρακαλώ, έχετε το λόγο. Κύριο Σιλικιώτης. Για την 33 ε, δεν ψηφίσαμε. Α, καταπίπτει. Καλώς. Εκτός μικροφώνου, πρόεδρος. Ψηφοφορία λοιπόν επί του συνόλου της ε, έκθεσης, ε, ονομαστική, πέραση ψηφοφορίας. Σαφές το αποτέλεσμα, εγκρίνεται τα συγχαρητήριά μας στον εισηγητή. Περνάμε λοιπόν εδώ τώρα στο σχέδιο γνωμοδότηση σε ό,τι αφορά την, μείωση, την ε, πρόταση οδηγία για τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον. Η κυρία Μπάρμπαρα Κάπελ είναι η συγγητριά μα. Συμβαστική ένα υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία ένα. Πέραση τη εγκρίνεται. 28. 85 Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 και 87 μαζί. Υπέρ, κατά, τις ελέγχουμε ηλεκτρονικά 86 και 87 λοιπόν. Από κοινού. Πέραση της φοβορίας. Εγκρίνεται. 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 89 υπέρ κατά να ελέγξουμε την 89. Πέραση της προφορίας εγκρίνεται. 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 91 απορρίπτεται 92 υπέρ κατά να ελέγξουμε και την 92 πέρασε απορρίπτεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να την αλλάξουμε και αυτή. 94 λοιπόν. Πέραση της φοφορίας, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 96 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 100 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 2α υπέρ Κατά. Ας ελέγξουμε. Συμβαστική τροπολογία 2α. Για να είμαστε απολύτως σίγουροι αφού πρόκειται για συμβαστική. Πέραση της φοφορίας. Εγκρίνεται. Εκατόν υπέρ. Κατά. Ξανά. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. απορρίπτονται 125, 126 και 127 από κοινού υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 128 υπέρ. Κατά. Για να την ελέγξουμε. Την 128 ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 129 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 130 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 131 υπέρ κατά για να την ελέγξουμε την 131 ηλεκτρονικά πέραση σφοφορίας Απορρίπτεται. 132 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε. 132. Πέραση της φοφορίας. Απορρίπτεται. Οι 133 και 134 καταπίπτουν, οπότε 135 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 136 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 137 υπέρ, κατά, για να ελέγξουμε την 137. Πέρασε της σφοφορία. Απορρίπτεται. 138 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 139 και 140 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Τις 139 και 140 από κοινού. Πέρασε τη Απορρίπτεται. Καταψηφίσατε κύριε. Καλώς. 141 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 142 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 144 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 145 υπέρ κατά ας ελέγξουμε την 145 πέραση της φοφορίας απορρίπτεται συμβαστική 3 υπέρ κατά να ελέγξουμε τη συμβαστική τροπολογία 3 είναι σημαντικό να την ελέγξουμε Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 152 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 153 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Και να σηκώνετε σας παρακολουθώ τα χέρια σας ε, όταν ψηφίζουμε, γιατί δεν σας βλέπω καλά. 153 λοιπόν, έχουμε Ψηφίζουμε τώρα ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε. Συμβαστική τροπολογία 4. Πέραση της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. έχουμε δύο τροπολογίες ως προσθήκες, 163 και 165. 163 καταρχήν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 ε, ε, λέω ο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ, Ας την ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τη σημασική τροπολογία 5. Πέραση στις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8 υπέρ. Κατά. Ελέγχουμε την τροπολογία 8. Ηλεκτρονικά λοιπόν. Πέρας. Απορρίπτεται λοιπόν 181 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Επαλήθευση της 181. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 182 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 184 υπέρ, κατά, επαλήθευση για την 184. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 185 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 186, 185, επαλήθευση λοιπόν για την 185. 185 πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Εξαιρετική ιδέα να το ελέγξουμε. 186 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την 186. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την 188. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε και αυτή. Ελέγχουμε την 189. Πέραση ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Κάντε την επιλογή σας. Πέρασε της ψηφορίας για τη συμβαστική τροπολογία 6. Εγκρίνεται. Ωραία. 205 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ. Κατά συγγνώμη, 210 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 209 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 212 υπέρ, κατά αποχές ε, απορρίπτεται, 213 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 214 υπέρ, κατά, να παληθεύσουμε τη 214. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Δεν έχει καμία σημασία ούτως ή άλλως. 215 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 217 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για τη 217. Επαληθεύουμε τη 217 πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 218 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 219 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 220 περ κατά, αποχές απορρίπτεται. 221 με 222 που είναι ταυτόσιμες υπέρ, κατά, επαλήθευση. 221 και 222. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 223. πάμε στη 242, κατά πάσα πιθανότητα στην ε, επόμενη σελίδα, τροπολογία του κυρίου Πάξας, τη 242, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 243 και 244, υπέρ, κατά, επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 245 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση και πάλι για τη 245. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 246 και 247 υπέρ, κατά, αποχές, να επαληθεύσουμε τη 246 και τη 247. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται. 248 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση και για αυτήν. 248. Δεν φαίνεται καθαρά το αποτέλεσμα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 249 περ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 250 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 251 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για τη 251. Πέρασε ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 252 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για τη 253. Καλύτερα να το επαληθεύσουμε και να είμαστε απόλυτα βέβαιοι. Πέραση της ψηφοφορίας. Είστε κατά? Απορρίπτεται λοιπόν η 253. 254 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε και πάλι. 254. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 255 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 256 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Γιατί δεν σηκώνετε τα χέρια σας. Δεν μπορώ να μαντέψω τι θέλετε να ψηφίσετε. 256, πέραση της ψηφοφορίας. Πέραση τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 257 υπέρ. Κατά. Σας παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας γιατί δεν καταλαβαίνω τίποτα. 2.57. Σας παρακαλώ. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Συγγνώμη. 2.57. Πέραση της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. 2.58. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 259 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 260 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 261 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 262 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 263 υπέρ κατά, απορρίπτεται, 264 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται, 265 υπέρ, κατά, αυτή τη φορά πρέπει να επαληθεύσουμε, 265, πέρασε της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 266 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 267 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται αυτή τη φορά. Συμβαστική τροπολογία 7 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για τη 17. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία 8. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Για την 27. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Για την 28. Ψηφίζουμε την 28. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, επαλήθευση Γιατί 37. Πέρα τη ψηφοφορία. Πώς ψηφίζετε, κύριε Βαμπρέντ, υπέρ, οπότε εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ, κατά. Εγκρίνεται, αλλά να κάνουμε και έναν ηλεκτρονικό έλεγχο καλύτερα. Συμβαστική τροπολογία 10 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρασε της ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για 42. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται από ό,τι αντιλαμβάνομαι. 43 υπέρ, κατά, επαλήθευση για τη 43. Πέραση της φορές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ, κατά, να ελέγξουμε τη 45. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 1 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Ελέγχουμε την τροπολογία 1. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 50, 50 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, 53 υπέρ, κατά, τώρα πρέπει να επαληθεύσουμε, 53. Πέρασε φορές ψηφοφορίες. Απορρίπτεται 54 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται, Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά τη συμβαστική τροπολογία 11. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12, ηλεκτρονικά και αυτή. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά πρέπει να την επαληθεύσουμε την 62 επαλήθευση για την 62 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται 63 υπέρ κατά επαλήθευση για την 63 πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 5 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά, επαλήθευση. 65. Πέραση ψηφοφορίας εγκρίνεται. 67 υπέρ, κατά. Να επαληθεύσουμε και την 67. πέρασε της ψηφοφορίες. Απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. 69. Επαλήθευση της 69. πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Που σημαίνει ότι πάμε στην 68. Υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 70 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται, 72 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 73 υπέρ, κατά, επαλήθευση για την 73, 73, πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 75 υπέρ, κατά, επαλήθευση για την 75. Πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται, 77 αποσύρεται, 76 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ, 76 μάλλον ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε της ψηφοφορίας, απορρίπτεται, 78 υπέρ, κατά, άποχες εγκρίνεται, 79 υπέρ, κατά, επαλήθεση για την 79. Επαλήθευση της 79, πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας και είμαστε και ακριβώς την ώρα μας. Τέσσερις και μισή. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Dear friends, uh... φίλη. Σύντομο διάλειμμα τριών λεπτών. Αν κάποιοι θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλώ ε, βγείτε το συντομότερο δυνατόν για να ξεκινήσουμε και χωρίς καθυστέρηση. Διακόπτουμε μόνο για τρία λεπτά. start Λοιπόν, σημείο 7 της σημερινής διάταξη υλοποίηση και λειτουργία του ονόματο τομέα ανωτέρου επίπεδου. EU. Ο Φεντρικ Φεντελίος συνάδελφο, καθίστερε από τον συνάδελφο Πέτερσεν εμπροκειμένο. Σας ευχαριστούμε. Όπως γνωρίζετε, το τελείο δημιουργήθηκε το 2002 με κανονισμό. Είναι καθιερωμένο, λειτουργεί ως όνομα το τα του επίπεδου, όμως το νομικό πλαίσιο πρέπει να ενημερωθεί για να έχουμε και το απαραίτητα ευέλικτο κανονιστικό περιβάλλον που χρειαζόμαστε. Προτείνει λοιπόν η Κομισιόν την καταργήση της υφιστάμενης νομοθεσίας. Οπότε, ε, συνάδελφε Πέτερσεν, παρακαλώ. Πρόεδρε, Ζητώ συγγνώμη εκ μέρους του κυρίου Φέντερλε, ο οποίος δυστυχώς αδυνατεί σήμερα λόγω κολλήματος. Η πρόταση είναι να καταργηθεί η τρέχουσα νομοθεσία, η φυσταμένη νομοθεσία. Θα συνεχίσει να λειτουργεί φυσικά το όνομα Όμως, πρέπει να προσαρμοστούμε στην ενομική πραγματικότητα και τις ανάγκες της αγοράς. Εν ώψη της ψηφιακής πολιτικής προσπαθούσαμε ανέκαθεν να λειτουργήσει καλά το .eu. Τα έχει καταφέρει, αλλά θέλουμε να συνεχιστεί αυτό και στο μέλλον, έτσι ώστε τα πλεονεκτήματα να ωφελήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συζητητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση και συμφωνεί ότι πρέπει να συνεχίσουμε να κινούμαστε δυναμικά στην αγορά ονομάτων τομέα και να είμαστε και ευέλικτοι. Η ύπαρξη του τελείου είναι πολύ σημαντική για την ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο συγητής πιστεύει ότι αποτελεί και μια ευκαιρία για θεσμούς, φορείς, οργανισμούς, εταιρείε να έχουν την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο όνομα του μένοντα του επίπεδου και αυτό βάσει κοινών κανόνων και αξιών. Η πρόταση θεσπίζει τους κανόνες καταχώρησης, θεσπίζει τα κρατηρία επιλεξιμότητας, τους όρους καταχώρησης και τους κανόνες αναστολής. Θεσπίζεται η σχετική νομοθεσία, η δυνατότητα κράτησης κάποιου ονόματος, καθώς και η διαδικασία διαπίστευση για τους καταχωρητέ ονομάτων. Στο κείμενο περιγράφονται λίγο πολύ τα πάντα, μεταξύ των οποίων και οι διαδικασίες όσον αφορά τις συμβάσεις με τους καταχωρητές. Εν γέννη, ο εισηγητής υποστηρίζει τη Γενική Αρχή. τονίζουμε στην ανάγκη να τονωθεί και να προβληθεί το .eu. Λαμβάνοντας υπόψη και την ανάγκη προστασίας κάθε λογής δικαιωμάτων. Εν ώψη των κανόνων του, του, κράτους δικαίου, ο εισηγητής ζητά επιπλέον εγγύησεις. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πιστεύουμε ότι πρέπει να προχωρήσουμε με κατεξουσιοδότηση πράξης. Υπάρχει ένα ζήτημα που χρήζει περαιτέρω συζήτηση και αυτό είναι το κατά πόσον ο χαρακτηρισμός του καταλόγου πρέπει να είναι στα χέρια μόνο μη κερδοσκοπικών επιχειρήσεων ή και κερδοσκοπικών. Κατά τη γνώμη του εισηγητή για ένα καλό κανονιστικό πλαίσιο, ένα καλό νομοθετικό πλαίσιο για να συνεχίσει να εμπλέκεται το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρέπει να θεσπίσουμε και εδώ τους σχετικούς κανόνες. Τέλος, ο εισηγητής ευχαριστεί την Κομισιόν, η οποία βοήθησε πάρα πολύ, απήντησε σε πολλές ερωτήσεις. Ο εισηγητής προσβλέπει σε περαιτέρω καλή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστεί και τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Συναδελφέ για την εισήγηση εκ του ΕΛΚ, ο κ. Χόπμαρ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τον συνάδελφο που παρουσίασε την έκθεση του ανταυτού. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε γρήγορα και εύκολα σε συμφωνία για να προχωρήσουμε με πνεύμα ρεαλιστικό. Με στόχο να βελτιώσουμε το 3U, το οποίο λειτουργεί ήδη πολύ καλά. Πιστεύω ότι ο σκοπός αυτού είναι η βελτίωση της εσωτερικής ψηφιακής αγοράς, η ενίσχυση της παρουσίας μας στο διαδίκτυο και η διευκόλυνση του διασυνοριακού εμπορίου. Ενώπιση δηλαδή και της ψηφιακής αγοράς. Μπορούμε λοιπόν να κάνουμε κάτι στο σημείο αυτό για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Θυμίζω ότι η νομοθεσία αυτή πρέπει να είναι απλή, να γραφούν ως δυνατόν περισσότεροι, αλλά και ασφαλής. Να παράσχουμε λοιπόν προστασία από hacker και άλλους που διαπράττουν έγνομες ενέργειες. Κάτι λοιπόν απλό και ασφαλές. Αυτές είναι οι δύο λέξεις κλειδιά. Καμιά φορά τα δύο αυτά ακούγονται αντιφατικά, γιατί για να είναι κάτι πολύ ασφαλές δεν θα είναι και απλό. Μπορούμε όμως να το περπηδήσουμε το εμπόδιο αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση να θυμάμαστε ότι υπάρχουν κανόνες και διαδικασίες. Και ας μην ξεχνούμε ποτέ την ανάγκη ασφαλείας, αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Θέλουμε το .eu να χρησιμοποιείται από αυτούς που έχουν δικαίωμα να το χρησιμοποιούν. Αυτά φυσικά λέγονται και στην πρόταση της Κομισιόν προς Ευρωπαίους πολίτες και ευρωπαϊκές εταιρείες, προς όσους ήδη επιχειρούν στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς όσους ε, έχουν οτιδήποτε συμφέρον από το .eu. Η προστασία, η, με συγχωρείτε, η πρόταση της Κομισιόν Ενέργεια είναι καλή. Έχουν κατατεθεί προτάσεις που νομίζω μπορούμε να υποστηρίξουμε, άλλε μπορούμε να τι συζητήσουμε. Προσβλέπω σε συζήτηση όσον αφορά την επίτευξη αυτού του διτού στόχου, όπως προείπα. Απλά και με ασφάλεια. Από τους σοσιαλιστές θέλει κανείς να πάρει το λόγο, παρακαλώ. θα μιλήσω εκ μέρους του κ. Τζορμαν και θα ήθελα να σα πω πως όπως έχει αναφερθεί ήδη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η λειτουργία ε, αυτού του ονόματος ε, τομέα ανωτά του επίπεδου από το 2005 έχει πραγματικά στεφθεί με επιτυχία και με βάση την ε, έκθεση αποτελεσμάτων ή επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει πράγματι ότι τα, οι στόχοι τους οποίους είχαμε θέσει παραμένουν οι ίδιοι. Αλλά υπάρχουν και νέες προκλήσεις στις οποίες θα πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά συνέπεια συμφωνούμε με τις προτάσεις του εισηγητή ε, ως προς ε, την τροποποίηση αυτή τη πρόταση τη ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ότι δηλαδή θα πρέπει, ε, είναι δικαιολογημένη μια τέτοια νέα πρόταση. Και πράγματι η αύξηση τη εμπιστοσύνη αποτελεί ένα από του βασικού στόχου. Ε, λαμβάνουμε υπόψη μα ότι η πρόταση τη Επιτροπή αποτελεί συνέχεια τη δημόσια διαβούλευση που έγινε τον Μάιο του 2017. Η συμπερίληψη των συνδυμάτων διακυβέρνηση μέσα στη νέα πρόταση είναι κάτι το πολύ ευπρόσδεκτο και υποστηρίζουμε τι προτάσει του εισηγητή για τροποποίηση τη πρόταση κανονισμού σε ό,τι αφορά ειδικότερα τα ζητήματα ε, ταυτότητα ε, του χρήστη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα δε στην ψηφιακή αγορά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, το... Η εφαρμογή των βασικών αρχών που θα αρχούν τα ζητήματα διακυβέρνηση του ε, ονόματο τομέα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των χρηστών είναι κάτι το οποίο είναι επίση ευπρόσδεκτο και θα πρέπει να το συζητήσουμε πέρα και με τον εισηγητή. Τώρα, ο ο στιώτης ε, ήρθε σε επαφή, μάλλον ήρθε σε επαφή μαζί του από την πλευρά ε, ενός IPO ε, και ε, πράγματι θα πρέπει να υποστηριχθεί η υποβολή αιτήσεων για την λήψη εμπορικών σημάτων μέσω των IPOs έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται σε αυτήν την κοινή ευρωπαϊκή ηλεκτρονική διεύθυνση. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θα προωθήσουμε περισσότερο το κοινό όνομα τομέα και με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να ε, καταπολεμήσουμε και καταχρηστική χρήση, για παράδειγμα, δηλαδή καταχωρήσει τέτοιων ε, domain names, δηλαδή ε, ονομάτων με αυτό το όνομα τομέα που δεν συμμορφώνονται με σχετικέ αρχέ. και επίση θα πρέπει να υπάρξει συμβολή υποστήριξη της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του κοινόμητρου. Ε, σε αυτή την ε, φάση βρισκόμαστε και σε φάση εσωτερική διαβούλευση από την πλευρά του σοσιαλιστέ και ε, ο συζητητέ μα θα διαβάσει την δηλαδή, δική μα θέση μόλι αυτή θα έχει οριστικοποιηθεί. Καλωσορίζουμε ε, λοιπόν την πρόταση από την πλευρά του εισηγητή. Αυτή λοιπόν ήταν η παρέμβαση του συνάδελφου. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Τσαβαρμένα λοιπόν ήταν, ε, τοποθετήθηκε εδώ Από την πλευρά τώρα του ECR, ο κύριο Στοσνόφσκι θα αντικαταστήσει τον κύριο Μπασίρ και θα πάρει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο συνάδελφο Μπασίρ μου ζήτησε να ζητήσω συγγνώμη εκ μέρου του και να διαβάσω την εξή δήλωση από την πλευρά του. και αισκιώδη λοιπόν συζητητή συμφωνεί με αυτή την πρόταση καθώς ε, το όνομα τομέα έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και στη μείωση του διοικητικού άχθους ε, σε ό,τι αφορά τους καταχωρητέ ειδικότερα. Ε, ο συνάδελφός μου θέλει να ευχαριστήσει τον εισηγητή για μια καλή πρόταση και υποστηρίζει τι περισσότερες από τις προτάσεις που κάνει. Παρότι συμφωνούμε ότι δεν θα πρέπει όλοι αυτομάτως να έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα τομέα.eu υπάρχουν ορισμένες ανησυχίες σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη πολιτικοποίηση του συζητήματος ε, όταν έχουμε να κάνουμε με την υποστήριξη των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ε, γνωστό ότι οι βρετανικέ, για παράδειγμα επιχειρήσεις ε, ενδέχεται να χάσουν το μέλλον την πρόσβαση που έχουν ακριβώ σε αυτή τη χρήση του νόματος ε, τομέα και γι' αυτό ο εισηγητή μα ε, θεωρεί πω θα πρέπει να βρεθεί μια λύση η οποία δεν θα θέσει σε ένα αμφιβόλο την ένθυμη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων και στο μέλλον και αναμένει ο συνάδελφο την συνεργασία με του υπόλοιπου εισηγητέ σε ό,τι αφορά αυτή την πρόταση που είναι τόσο σημαντική για την κοινή αγορά. Ευχαριστώ, Λέω Δεν υπάρχει κάποιο άλλο που να θέλει να πάρει το λόγο. Οπότε θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκρίνια από τη Γενική Διευθύνση Connect για να τοποθετηθεί εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Φέντελε για αυτή την θετική εκθεσή του και για την συνεργασία που είχαμε στο πλαίσιο της σύνταξης αυτής της έκθεσης. Όπως αναφέρθηκε ήδη, έχει ξεκινήσει εδώ και 12 χρόνια ήδη αυτό το όνομα τομέα, η EU, προκειμένου να προωθήσουμε μια κοινή ονομασία στο διαδίκτυο και έχει σχεδιαστεί για να προωθήσει τις κοινέ αξίες, αλλά και να παρέχει περισσότερη εμπιστοσύνη στους χρήστες σε ό,τι αφορά τη σταθερότητα και την αξιοπιστία του ιστοτόπου. Και πράγματι, αυτό καταδεικνύει από το γεγονό ότι σήμερα έχουμε 3,8 εκατομμύρια καταχωρήσει υπό αυτό το όνομα τομέα. Η πρόταση τώρα στοχεύει στον εξυγχρονισμό του ε, νομοθετικού πλαισίου μέσω μια ε, πιο ελαφριά εντό εισαγωγικών και προσανατολισμένη στι αξίε μα ε, διαδικασία καταχώρηση και μια, διαδικασία η οποία παρέχει περισσότερη καταχώρηση, ευελιξία προκειμένου να γίνεται και κατάλληλη προσαρμογή στι νέε εξελίξει στον τομέα τη βιομηχανία των ομάδων τομέα. Επίση, η νέα πρόταση βελτιώνει διακυβέρνηση μέσω της δημιουργίας ενός ε, συμβουλευτικού συμβουλίου από διάφορους τομείς, ε, συμμετέχοντες δηλαδή από, τους, ε, από τα κράτη-μέλη, από την Ένωση, από τους ενδιαφερόμενους εφορείς, ε, αλλά και από την οικονομική κοινότητα, έτσι ώστε όλοι να έχουν το δικό τους λόγο σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του ονόματος στο τομέα, ακολουθώντας την ίδια συλλογιστική που ακολουθούμε σε ό,τι αφορά τη κυβέρνηση του διαδικτύου. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω πως η νέα πρόταση διευρύνει το δικαίωμα καταχώρηση υπό αυτή την ονομασία ε, στους ε, πολίτε Ευρωπαϊκή Ένωση που διαμένουν σε άλλε χώρε. Δηλαδή, οι πολίτε αυτοί θα είναι πλέον σε θέση να συνδέονται χρησιμοποιώντα την δική του ευρωπαϊκή online ταυτότητα όπου και βρίσκονται στον κόσμο. Ο βασικό μα στόχο είναι να δούμε περισσότερου ανθρώπου και περισσότερε επιχειρήσει να χρησιμοποιούν αυτό το όνομα τομέα προκειμένου να συμμετάσχουν περισσότερο στην ε, κοινή ψηφιακή αγορά και προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να δώσουν το στίγμα, αν θέλετε, τη ευρωπαϊκή του ταυτότητα online, αλλά και προωθώντα τι ευρωπαϊκέ αρχέ σε ό,τι αφορά την πολυγλωσία, την προστασία τη προσωπική ζωή, αλλά και την ασφάλεια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Φέντελε, να σας δώσω, ή ε, μάλλον κύριε Πέτερσεν που αντικαταστάτε τον κύριο Φέντελε για να πείτε δύο λόγια, γιατί αφού αντικαταστάτε τον εισηγητή θα πρέπει να πείτε δύο λόγια. Ναι, Πρόεδρε, είναι εύκολο να το κάνω γιατί έγιναν πολλά επικοδομητικά σχόλια και είμαι σίγουρος ότι ο εισηγητή θα είναι ευγνώμων για όλα αυτά τα σχόλια και ότι αναμένει με ενδιαφέρον τη συνεργασία με του υπόλοιπου αισιώδει εισηγητέ. Αντιλαμβάνομαι ότι ο στόχο του είναι να έχουμε καταλήξει από αυτού του φακέλου έω τα τέλη αυτού του χρόνου, πράγμα το οποίο δείχνει να είναι πραγματικά πάρα πολύ πιθανό βασιζόμενο στα σχόλια που ακούστηκα σήμερα Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πέτερσεν. Περνάμε τώρα σε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις. 26 Νοεμβρίου 2018 είναι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών ε, ψηφοφορία στην Ήτρε στις 26 Σεπτεμβρίου, συγγνώμη, ψηφοφορία στην Επιτροπή 21 Νοεμβρίου. Επόμενο θέμα, προώθηση της δικαιοσύνης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες των διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Πολύ σημαντικό θέμα, η διαμεσολάβηση και οι υπηρεσίες αυτές. Υπάρχει γνωμοδότηση βάσει του άρθρου 53 προς την ΙΜΚΟ που είναι η αρμόδια επί της ουσίας ε, ε, επιτροπή. Θα ήθελα να ε, δώσω στο λόγο στη συντάκτρια της γνωμοδότησης, την κυρία Ζαμπόρσκα, για να μιλήσει πρώτη. Παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Βάσει αυτό του σχεδίου κανονισμού για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες διαδικτυακών υπηρεσιών διαμεσολάβησης είναι δύο πράγματα. Πρώτον, οι διάφοροι τρόποι των καθημερινών ε, επαφών μεταξύ των επιχειρηματικών χρηστών και των υπηρεσιών διαμεσολάβησης ή μεταξύ των χρηστών με τις ιστοσελίδες τους και τις ε, μηχανές αναζήτησης ε, αφετέρου. Πρόκειται για τα άρθρα 3 έως 8 του προτιμνόμενου σχεδίου. Εδώ αναφερόμαστε στις επιχειρηματικές συνθήκες, την διακοπή των υπηρεσιών, τους κανόνες ταξινόμησης, καθώς επίσης και τους ε, ε, κανόνες ίσης μεταχείρισης, ε, πρόσβασης ε, και της δυνατότητας να προσφέρονται διαφορετικές προϋποθέσεις με διάφορα μέσα. Υπάρχει και μία πληθώρα άλλων θεμάτων που αφορά την επίλυση διαφορών στα άρθρα 9 ως 12 και έχουμε και αντίστοιχε συνθήκες ε, για τα συστήματα μεταξύ της κάθε πλατφόρμες για την επίλυση των καταγγελιών. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιείται η υπηρεσία διαμεσολάβησης και επίσης δημιουργείται και πεδίο για ε, ομαδικές αγωγές. Όπως γνωρίζετε, η Επιτροπή μας, η Ήτρε, έχει ενισχυμένες αρμοδιότητες για τα άρθρα 5 και 6 που αναφέρονται στην ταξινόμηση και στην άνηση ή διαφορετική μεταχείριση. Σε γενικές γραμμές, το σχέδιο κειμένου που μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι αρκετά ποιοτικό, είναι ένα ισορροπημένο έγγραφο ε, πολλοί το επικρίνουν, αλλά για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, επομένως εγώ θεωρώ ότι είναι ισορροπημένο. Και η πρόταση που έχω εγώ στο έγγραφο είναι ένα συνδυασμό μιας φιλόδοξης προσέγγισης, ε, διότι θεωρώ ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε κάποια σημεία παρά είναι προσεκτική και κάποια άλλα σημεία στα οποία θεωρώ ότι η πρόταση είναι πολύ φιλόδοξη όσον αφορά την παρούσα ε, λειτουργία του ψηφιακού οικοσυστήματος. Ε, γνωρίζω και το σχέδιο έκθεσης τώρα της ε, στην Επιτροπή ΙΜΚΟ. Νομίζω ότι δεν θα έχει πρόβλημα με τα δικά μου σχόλια και φυσικά ε, περιμένω και τις τροπολογίες σας. Νομίζω ότι κάνω δύο φιλόδοξες προτάσεις. Καταρχάς θα ήθελα το νέο έγγραφο, ο νέος κανονισμός να καθορίζει υποχρεώσει για τι πλατφόρμε και τι μηχανέ αναζήτηση για να προσφέρουν πρόσβαση σε δεδομένα σε επιχειρηματικού χρήστε και ιστοσελίδε, δεδομένα τα οποία παρέρχονται από τι αμοιβέ συναλλαγέ μεταξύ πλατφόρμα και επιχειρηματικού χρήστη και καταναλωτή. Αλλιώ ε, επιτρέπουμε στι πλατφόρμε και στι μηχανέ αναζήτηση να ιδιωτικοποιούν δεδομένα τα οποία δεν θα έπρεπε να ε, χρησιμοποιούν ε, με αποκλειστικά δικαιώματα. Και επίση θεωρώ ότι πρέπει να απαγορευτεί ε, η πρακτική που χρησιμοποιούν κάποιε υπηρεσίε διαμεσολάβηση που περιορίζουν τα δικαιώματα εμπορικών επιχειρηματικών χρηστών να παρέχουν ε, μέσω άλλων διάβλων τις ίδιες υπηρεσίες και τα ίδια προϊόντα με πιο προνομαϊκές συνθήκες, γιατί αυτό ε, περιορίζει το, την ελευθερία του επιχειρήν και θα δημιουργήσει πρόβλημα στο νομοθετικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης αργά ή γρήγορα. Ολοκληρώνω ε, με τη θέση μου για κάποια θέματα τα οποία θεωρώ ότι είναι η ενισχυμένη μας αρμοδιότητα της Επιτροπής μας. Όσον αφορά την ταξινόμηση, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, υπερβαίνει λίγο τα όρια και το θέμα της διαφάνειας ε, της ταξινόμησης θα πρέπει να αφορά τις παραμέτρους και όχι τους λόγους για τους οποίους έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες παράμετροι και όχι κάποιες άλλες, διότι ορισμένες φορές δεν μπορεί να δώσει κάποιο μια λογική εξήγηση γιατί ο καταναλωτής συμπεριφέρεται με κάποιο τρόπο και αυτές οι παράμετροι έχουν περιγραφικό και όχι ε, αφηρημένο χαρακτήρο. Και επίσης να σας πω και κάτι Όσον αφορά την άνηση μεταχείριση, αποφάσισα να συμπεριλάβω και τις υπηρεσίες αναζήτησης στον τομέα αυτό. Σήμερα το συζητήσαμε με εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι μας είπαν ότι όσον αφορά τις ε, μεγαλύτερες μηχανές αναζήτησης, υπάρχει ήδη απόφαση για απαγόρευση τέτοια συμπεριφορά ε, και αν υπάρχει υποχρέωση ενημέρωση για διαφορετική μεταχείριση όσον αφορά ε, την αναζήτηση, ε, μπορεί αυτό να ε, ερμηνευθεί ως ανοχή αυτής της συμπεριφοράς αρκεί να είναι διάφανη όλη η διαδικασία. Αυτό είναι εύλογο επιχείρημα και θα το εξετάσω προς το παρόν. Δεν μπορώ να σας πω κατά πόσον συμφωνώ ή διαφωνώ με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ευχαριστώ πολύ. Α, είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, κύριε Ζωρινιό, αντικαθιστάτε την κυρία Καηλή από τους σοσιαλιστές. Παρακαλώ. Πρόεδρε, η συναδελφός μου Εύα Καηλή ζητά συγγνώμη, δεν μπορεί να περαστεί. Εκπροσωπεί όμως το Κοινοβούλιο σε συνέδριο στις ΗΠΑ. Ευχαριστούμε την Κομισιόν για την αρχική της πρόταση και τον εισηγητή για το έργο του, τη μελέτη του φακέλου. Πολύ σημαντική νομοθετική πράξη αφορά την επόμενη εντολή αλλά και τα επόμενα χρόνια. Η ΙΤΡΕ ενδιαφέρεται εκ των πραγμάτων για να προστατεύσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να μην σταματήσουμε την καινοτομία θέτουμε τις προποθέσεις για διαφάνεια και προσβλέπουμε στα επόμενα βήματα. Ταυτόχρονα θέλουμε να προστατεύσουμε τις επιχειρήσεις από την αυθαίρετη διακοπή παροχής τέτοιων υπηρεσιών. Επίσης, προσπαθούμε να σταματήσουμε παράνομο περιεχόμενο. Οι κανόνες κατάταξης επίσης ε, πρέπει να είναι διαφανή και εύκολα κατανοητή. Πρέπει επίση να διευκολύνουμε την προστική φωνής και εικόνας. Θέλουμε ισότιμη μεταχείριση όλων των αγαθών και υπηρεσιών. Όπως είπα, χρειαζόμαστε διαφάνεια, περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση των καταναλωτών. Η Εύμα λοιπόν μου ζήτησε να σας μεταφέρω ότι προσβλέπει και σε μια επικοδομητική διαδικασία επίλυσης διαφορών και είναι βέβαιο ότι θα εξευρεθεί μια τελική λύση. Επί Τετάρτη λίγη προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών πρέπει να συνεργαστούμε τάχιστα. Εκ μέρους της Εύας Καηλή, ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή και θα συζητήσει φυσικά τις συμβαστικέ τροπολογίες, κατά το οποίο θα μας επιτρέψει να κλείσουμε το θέμα για τα ευρωπαϊκά όργανα. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε, λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστώ για την αντικατάσταση της ε, σκιώδωσή του. Οπότε, η κυρία Φίρινγκ, που αντικαθιστά την κυρία Λίνα. Πρόεδρε, οι επιγραμμικές πλατφόρμες όπως οι μηχανές αναζήτησης, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή ηλεκτρονικού δικτύου έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο που κάνουμε τις αγορές μας. Διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους επενδυτές και ικανοποιούν καλύτερα τις ανάγκες των καταναλωτών. Σήμερα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής την ενιαία ψηφιακή αγορά. Κάνουμε ένα βήμα για να διευκολύνουμε τις επιχειρήσεις οι οποίες επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν μέσω πλατφορμών στην εσωτερική ψηφιακή αγορά. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το κείμενο που τονίζει ότι ο στόχος μας είναι να επιτρέψουμε τους παράγοντες της αγοράς να προχωρήσουν μέσα σε κλίμα διαφάνειας. Ο κανονισμός είναι οριζόντιος πολιτεομεακού ενδιαφέροντος. Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε ότι όλοι εκπροσωπούνται εξίσου και ισότιμα σε όλες τις πλευρές. Όχι λοιπόν στα περί τα εμπόδια και στις τρευλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται είτε επιγραμμικά είτε φυσικά στην αγορά. Να προσέξουμε επίσης οι επιγραμμικές πλατφόρμες και οι μηχανές αναζήτησης πρέπει να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες όταν λειτουργούν για τον ίδιο σκοπό. Δεύτερον, αυτή είναι τη στιγμή οι πάροχοι υπηρεσιών αναζήτησης πρέπει να φροντίζουν να ισχύουν ίδιοι κανόνες για όλους. Όλους τους παρόχους αγαθών ή υπηρεσιών, είτε όταν αυτό γίνεται αμέσως είτε εμέσως είτε υπάρχει έλεγχο στο περιεχόμενο δηλαδή, είτε όχι. Μια καλύτερη λοιπόν πιο ισορροπή προσέγγιση στις υπηρεσίες διαμεσολάβηση μεταξύ πλατφορμών και πολιτών. Εκεί χρειάζεται ισοτιμία. Οι επαγγελματίες χρήστες πρέπει επίσης να έχουν το την δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στα στοιχεία τους και στα στοιχεία των συλλαγών για να είναι σε θέση να αναβαθμίσουν τα συστήματά τους και να παρέχουν εξαιρετικές υπηρεσίε στους χρήστες τους. Τέλος, πρέπει να εξετάσουμε τους παράγοντες και τα κριτήρια κατάταξης, γιατί έτσι μόνο θα υπάρξει διαφάνεια και δικαιοσύνη, αλλά και εν τέλει δίκαιος ανταγωνισμός, χωρίς να αποκαλύπτουν οι ή οι δε κάποια εμπορικά τους μυστικά. Όσον αφορά το σύστημα επεξεργασίας παραπώνων, πρέπει όντω να παραπέμπονται στην καθετερία σε του μεγέθους της. Επίσης, με βάση αυτά, οι πελάτες, οι καταναλωτές αλλά και οι επενδυτές θα μπορούν να λάβουν αποφάσεις με τα λόγου γνώσεως. Κύριε θα υποβάλει συμβαστικές τροπολογίες και να αυτού ε, προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία. Ευχαριστώ. Και ο Σάκερβολ από την Επιτροπή και δει την Γενική Διεύθυνση Connect. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την κυρία Σιγητή. Ε, καταρχήν να σας αναφέρω πως η DigiConnect και η DigiGrowth ε, ε, συνεργάζονται από αυτού του φαγγέλου και καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τα μέλη εδώ της Επιτροπής σας ε, για το γεγονός ότι αντιλαμβάνονται τα περίπλοκα ζητήματα ε, αυτού του φακέλου ε, τα οποία προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε εμείς με την πρότασή μας και πραγματικά επιχαίρουμε το γεγονός ότι έχετε κατανοήσει επακριβώς το τι ακριβώς προσπαθούμε να κάνουμε και το ακούσαμε αυτό από όλες τις παρεμβάσεις και ειδικότερα μέσα στην πρόταση της Ιρία Ζαμπρόσκα. Επιτρέψτε μου να εξηγήσω καταρχήν ότι η στη λογιστική ε, πίσω από την πρόταση παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι θα πρέπει να ε, λάβουμε κάποια σημαντικά και άμεσα μέτρα ε, για να αντιμετωπίσουμε τις περιπτώσεις εκείνες όπου υπάρχουν καταχρηστικές συμπεριφορές ή αδιαφανείς συμπεριφορές παράτυπες και γνωρίζουμε ε, φυσικά ότι υπάρχουν βασικές αρχές διαφάνειας ε, ε, που διέπουν την πρόταση. Και εκείνο βέβαια που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και για αυτή την Επιτροπή είναι η δυνατότητα πρόσβαση σε τέτοιου είδου υπηρεσίες διαμεσολάβηση αλλά αυτό και το, το νέο δικαίωμα που υπάρχει για τις ομαδικές ε, προσφυγές ε, σε ό,τι αφορά για παράδειγμα ομοσπονδίες ε, επιχειρήσεων. Αυτές λοιπόν οι δυνατότητες δίνουν άμεσες δυνατότητες προσφυγής για μικρού μεγέθους επιχειρήσεις οι οποίες δηλαδή βασίζονται ακριβώς σε αυτές τις online πλατφόρμες διαμεσολάβησης και χωρίς αυτές δεν ξέρουν σε ποιον απευθυνθούν, δεν έχουν σε ποιον απευθυνθούν. Ένα δεύτερο ζήτημα που θα ήθελα να αναφέρω και το οποίο ήδη αναφέρθηκε εδώ είναι το ότι υπάρχουν μία σειρά από περιπτώσεις για τις οποίες ε, δεν μπορούσαμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι ήταν απαραίτητε σε πιο αυστηρέ ε, απαγορεύσει ή μέτρα, για παράδειγμα σε ό,τι αφορά την ε, πρόσβαση σχετικέ πληροφορίε ή τι ρήτρε τύπου Πρασπάρτη. Οπότε προστείνουμε καταρχήν κάποιε διατάξει ό,τι αφορά τη διαφάνεια και αποκοινούμε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, το οποίο θα συνέλθει μάλιστα για πρώτη φορά στα, αργότερα μέσα σε αυτή την εβδομάδα. Αποφασίσαμε να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση προκειμένου να αντλήσουμε κάποια συμπεράσματα ω προ το κατά πόσο είναι αναγκαία ε, κάποια επιπρόσθετα μέτρα στο μέλλον. Επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια σε σχέση ε, με κάποιε από τι βασικέ τροπολογίε που προτείνει η κυρία Ε, είπε ήδη η ίδια, και εμεί κατά την προετοιμασία τη πρότασή μα, είχαμε αναλογιστεί ε, κάποιες από αυτέ τι δυνατότητε που προτείνει, για παράδειγμα, επέκταση του άρθρου 6 και σε ό,τι αφορά το άρθρο 7, δηλαδή τι ε, ε, διαδικτυακές αναζητήσεις, αλλά θεωρήσαμε ότι τέτοιου είδου προτάσει θα πήγαιναν ε, πολύ μακριά ειδικότερα σε ό,τι αφορά τον ευρύ ε, και συμμετοχικό χαρακτήρα αυτού του εργαλείου. Γιατί, όπω γνωρίζετε, με βάση την αξιολόγηση αντικτύπου υπάρχουν 7.000 ε, τέτοιου είδους ε, μικροπλατφόρμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, ε, σε σχέση με τις περαιτέρω προτάσεις, θα θέλω να σας πω ότι αυτή την περίοδο εμείς από την πλευρά της Επιτροπής βρισκόμαστε σε μια φάση παρακολούθησης προκειμένου να διαπιστώσουμε σε ποιο βαθμό έχουν υπάρξει αποτελεσματικέ οι που θεσπίστηκαν από ορισμένα κράτη-μέλη. Αυτά από την πλευρά μου και φυσικά είμαστε στη διάθεσή σα για περαιτέρω ανταλλαγέ απόψεων ε, στο πλαίσιο δηλαδή τη περαιτέρω εξέταση αυτού του φακέλου από την πλευρά τη Επιτροπή. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Ε, η συγγήτριά μα έχει και πάλι το λόγο για τα καταλητικά σχόλια, κυρία Ζαμπόρσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ θερμά του συναδελφού ε, Ζώνη και Φίρινγκ που παρουσίασαν τις τοποθετήσεις εδώ των σχεδόν εισηγητών, αλλά και ευχαριστώ και την Επιτροπή για τα σχόλια της. Ε, νομίζω πως ε, τα όσα ακούστηκαν σήμερα εδώ καταδεικνύουν ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερες διαφορές απόψεων σε σχέση με αυτό το θέμα. σε ό,τι αφορά δηλαδή την, την τοποθέτηση από την πλευρά αυτή εδώ τη Επιτροπή Ήτρε. Οπότε αναμένω με ενδιαφέρον την περαιτέρω συζήτηση και τι τροπολογίε που θα υποβάλουν οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ, λέει ο συνάδελφο. «26 Σεπτεμβρίου είναι η προθεσμία, έτσι, στις 12 το μεσημέρι, Τετάρτη, λοιπόν για την υποβολή των ε, τροπολογιών, δηλαδή σε δύο μέρες, σε λιγότερο από δύο μέρες, έτσι. Και μετά στις 6 Δεκεμβρίου στην ΙΜΚΟ θα γίνει η ε, τελική ψηφοφορία. Επόμενο λοιπόν είναι σημείο, τεχνολογία blockchain, μια μακρόπνοη εμπορική πολιτική. Μία έκθεση λοιπόν πρωτοβουλίας και στο πλαίσιο του άρθρου 54 χρειάζεται και τοποθέτηση από τη δική μας πλευρά. Και να σας πω ότι εδώ τα ζητήματα, τα τεχνολογικά αλλά και τα ζητήματα καινοτομία σε σχέση με αυτές τις τεχνολογίες distributed ledger ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την Επιτροπή μας και έχουμε ήδη ε, συζητήσει αυτό το ζήτημα και είχε υπάρξει και ένα ψήφισμα από την πλευρά μας το 2018 ε, και στο παρελθόν μας απασχόλησε επανειλημμένα αυτό το ζήτημα στο πλαίσιο διαφόρων προτάσεων και θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο ε, στον ε, εισηγητή μας, τον κύριο Κρίσταν Σίλβιο Μπουσόε να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι το μέλλον της ανταγωνιστικότητας και της δυνατότητας καινοτομίας ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να σχετίζεται στενά με την ε, έγκριση και διανομή των λεγόμενων DLT, των Distributed Ledger Technologies. Ε, επίσης, μπορεί να υπάρχει σχετική διαμόρφωση της βιομηχανίας μέσω αυτών των ε, νέων τεχνολογιών. Έτσι μπορούμε να έχουμε καλύτερα εμπορικά συστήματα μέσω διάφανων συνθήκων, να μειωθεί το κόστος επιμελητίας με πολύ σημαντική μείωση σε τεκμηρίωση και κόστος επαλήθευσης, ε, μείωση της γραφειοκρατίας, αύξηση της ασφάλειας, προστασία των καταναλωτών και κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τα κριτήρια λήψης αποφάσεων. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης Επιτροπής μας, προσπάθησα να είμαι όσο το δυνατόν πιο λακωνικός, αλλά να συμπεριλάβω και τα πάντα. Ήμουνα σε στενή επαφή με τους σκιώδεις συντάκτες και του συμβούλους μας και τα βασικά σημεία στα οποία επικεντρώθηκα στη γνωμοδότησή μου είναι τα εξή. Η έκθεση της ΣΥΝΤΑ αναφέρεται σε συγκεκριμένο τρόπο DLT, σε τύπο DLT, ε, που είναι το blockchain ε, με ιδιωτική άδεια. Εγώ θέλησα να επικεντρωθώ και σε νέες μορφές ε, DLTs, οι οποίες ακόμα είναι σε εξέλιξη. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα οικοσύστημα ε, στο οποίο οι νεοφυείς επιχειρήσεις ε, θα ευνοούνται και θα υπάρχει πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Ζητώ επίσης ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κρατών μελών για να χρησιμοποιούνται αυτές τις τεχνολογίες για να βελτιώσουμε την παρακολούθηση, την ασφάλεια και το μηχανισμών επαλήθευσης για να καταπολεμήσουμε παράνομες πληρωμής, ε, να ε, δημιουργήσουμε προβλήματα για το ξέπλυμα χρήματος και να μπορούμε να προστατεύσουμε στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες εφαρμογές για τις ε, διαδικασίες διεθνούς εμπορίου, αλλά ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως η τεχνολογία ώστε να μπορεί να θεωρείται ότι μπορεί να εφαρμοστεί από νομική σκοπιά. Όσον αφορά τις συνέπειες για το πυρεβάλλον, ε, οι DLTs γενικά και οι μηχανισμοί συνένωση blockchain θα πρέπει να είναι φιλικοί προς το περιβάλλον και να μην είναι τόσο ενεργοβόροι. Ανέφερα επίσης ότι υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τεχνολογίες αυτές ε, μαζί με άλλες τεχνολογίες όπως το ίντερνετ των πραγμάτων, ε, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. και να ε, μελετήσουμε περαιτέρω τη δυνατότητα να υπάρχει ψηφιακή μετατροπή. Και ένταξη στο διεθνές εμπόριο. Αναφέρθηκα επίσης στις δυνατότητες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δει προκλήσεις ασφαλείας, να αξιολογήσει ε, κινδύνους και να υπάρξουν μέτρα για να αντιμετωπίσει αυτούς του κινδύνους. Όσον αφορά τους ε, ε, κβαντικούς υπολογιστέ, προτείνω να προχωρήσουμε τα θέματα αυτά. Επίσης, ε, καλωσορίζω ε, τη δουλειά που κάνει το EU Blockchain and Observatory Forum και ενθαρρύνω τη μελέτη εφαρμογών για να διευκολύνει το διεθνές εμπόριο. Ε, έχουμε μια εταιρική σύμπραξη που περιλαμβάνει 25 κράτη-μέλη και την Νορβηγία και θεωρώ ότι είναι πολύ καλός τρόπος για να εξετάσουμε τους μελλοντικούς τομείς σε θέματα κανονιστικά. Επειδή υπάρχει περιορισμός ε, στις ε, ε λέξεις που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη γνωμοδότηση. Σας παρακαλώ να στείλετε τις τροπολογίες σας στα αγγλικά, γιατί αύριο λίγη ε, προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Προσβλέπω στην συνεργασία και περιμένω και τις συμβαστικές τροπολογίες μέχρι την ημερομηνία. Η κυρία Βίρινγκ είναι σκιώδηση συγγήτρια εξ ονόματος των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουσόη για το σχέδιο γνωμοδότησης και για το γεγονός ότι ήδη έλαβε υπόψη του κάποιες προτάσεις των φιλελευθέρων. Θα σταθώ σε τρία στοιχεία τα οποία ακόμα δεν έχει θίξει ο εισηγητή κατά την άποψή μου. Πρώτον, είναι γεγονό ότι το blockchain δεν είναι μια εφαρμογή, αλλά η τεχνολογία η οποία διέπει πολλέ νέε εφαρμογέ. Άρα θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να υπάρξει νομοθεσία για τις εφαρμογές. Ιδάλλως, ε, θεωρώ ότι περιορίζουμε την καινοτομία και τη δημιουργία νέων εφαρμογών. Δεύτερη παρατήρηση, οι ευκαιρίες που προσφέρει το blockchain για τις ενεργειακές αγορές. Όταν θα αρχίσει η εφαρμογή αυτής της νέας τεχνολογίας θα βρισκόμαστε ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το blockchain μπορεί να βοηθήσει τις ενεργειακές αγοράς παρέχοντας ε, αυτόματα έξυπνα συμβόλαια με χρήστες που θα έχουν αυτή τη δυνατότητα. Και τελευταία παρατήρηση για την επανάσταση που ε, προϋποθέτει αυτή η νέα τεχνολογία για τον ε, κλάδο, τους ενδιαφερομένους και τους εργαζομένους. Θα πρέπει να δούμε τι αντίκτυπος θα υπάρχει για όλους τους τομείς. Αυτή η νέα τεχνολογία θα μπορούσε να επιλύσει και λεπτά ζητήματα όπως ε, θέματα πνευματικών δικαιωμάτων. Ιδίω την ανάπτυξη έξυπνων πνευματικών δικαιωμάτων που θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα καταθέσω σχετικέ τροπολογίες και προσβλέπω στη συζήτηση στις του των Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Καϊλή αυτή τη φορά εκπροσωπείται από τον κύριο Νίκα. Ευχαριστώ. Ζητά συγγνώμη κύριε Καϊλή. Κολλείεται όμως. Θα κάνω ότι μπορώ να μεταφέρω το μήνυμά της. Η κυρία Καϊλή εκφράζει την ικανοποίησή τη για την γνωμοδότηση υπέρ του Διεθνούς Εμπορίου. Ξεκίνησε με ένα ψήφισμα για το blockchain που θα ψηφιστεί τον Οκτώβριο. Η πρόταση της ΙΝΤΑ ανήκατοπτρίζει και τη δική μας θέση. Πρόκειται για ένα πλαίσιο υπέρ της νέας τεχνολογίας για να εξασφαλίσει ουδετερότητα στις συναλλαγές. Αυτές οι τεχνολογίες ε, καταχώρηση επιτρέπουν και τη λειτουργία του blockchain. Για μας δεν πρόκειται μόνο για την εφαρμογή, πρόκειται για υποδομές πολύ σημαντικές διαμεσολαβούντων συστημάτων μεταξύ διαφορετικών αρχείων καταχώρησης θα εγκαταστήσουν από ό,τι φαίνεται πολλά παραδοσιακά συστήματα. Αυτά θα αυτοματοποιήσουν το διεθνές εμπόριο σε πολύ μεγάλο βαθμό. Η Κομισιόν καλείται συναφώς να εξετάσει το θέμα. Η Κομισιόν πρέπει να συνεχίσει την έρευνα για το blockchain για να μειωθεί η φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή και να ελέγχονται πληρωμές. Φυσικά υπάρχουν και ανησυχίες όσον αφορά την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, σε αυτό το νέο περιβάλλον. Χρειάζεται και συμμόρφωση με τον GDPR και προστασία γενικότερα των προσωπικών δεδομένων. Το blockchain δημιουργεί νέες προοπτικές για να αφήσει επιχειρήσεις αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλο το μήκος της αλυσίδα εφοδιασμού. Θα δούμε πως το blockchain και οι σχετικές εφαρμογές θα οδηγήσουν σε έξυπνες πληρωμές ποιότητα και αξιοπιστία στις πληρωμές και τις συναλλαγές γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας και ευχαριστώ που μου δώσατε την δυνατότητα να μιλήσω εκ μέρους της κυρίας Καΐλη. Πρόεδρος. Χαίρομαστε πολύ που η κυρία Καΐλη μίλησε εξ ονόματός σας από την Κομισιόν, ο κ. Σάγκεβολ και πάλι από την Γενική Διεύθυνση Connect. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ τον ισχύτη και πάλι συγχαρητήρια, εξαιρετική έκθεση. Δύο παρατηρήσεις μόνο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακολουθεί το κοινοβουλίο που ήταν πρωτοπόρο στον τομέα, να γνωρίσει την αξία της τεχνολογίας και χαιρόμαστε που σε αυτήν την Επιτροπή για άλλη μια φορά γνωρίζετε η σημασία της τεχνολογίας. Η Ευρώπη πρέπει να είναι στο προσκήνιο πρωτοπόρος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συναφώς δημιούργησε ένα παρατηρητήριο για το blockchain καθώς και ένα αντίστοιχο φόρουμ στο οποίο συμμετέχουν πολλά κράτη-μέλη. Το παρατηρητήριο μελετά διάφορες περιπτώσεις, καταγράφει πρωτοβουλίες που εκδηλώνονται εδώ και εκεί σε μικρό αριθμό πλατφορμών, κυρίως των ευρωπαϊκών βεβαίως, όπου αρχίζει να διαφαίνεται το δυναμικό που διαμορφώνεται. Σημειώνουμε τις προτάσεις να μελετήσουμε τις εφαρμογές που διευκολύνουν το διεθνές εμπόριο. Ακόμη δεν είναι από τις υψηλές προτεραιότητές μας, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες συναντήσεις, πάντως προσβλέπουμε στην έκδοση της γνώμης του Κοινοβουλίου και από εκεί πέρα εννοείται θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βοηθήσουμε την Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και για να κλείσουμε, ο εισηγητής μας, ο κ. Φουσόη. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Γιάννη και την κυρία Καηλή και τον Σάλφα Τενίκα βεβαίω. Ε, νομίζω ότι όλοι συγκλίνουμε προς αυτά που είπα και εγώ. Το κείμενο πάντως μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Το θέμα είναι να στείλουμε ένα σαφές σήμα, ένα σαφές μήνυμα ότι πρέπει να είμαστε πρωτοπόροι στην τεχνολογία. Πρέπει να υποστηρίζουμε αυτή τη διαδικασία και φυσικά παράλληλα πρέπει να υπογραμμίζουμε τους κινδύνους. Διότι δηλαδή, εδώ, αν προκειμένου, έχουμε να κάνουμε μια τεράστια ευκαιρία για την βιομηχανία να γίνει πιο ανταγωνιστική. Αναμένω τροπολογίες και δεσμεύομαι ότι θα συντάξω ως το δυνατόν περισσότερες συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους. Πρόεδρος. 8 Οκτωβρίου 18, 6 το απόγευμα είναι η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. 10 μέρες δηλαδή από σήμερα. Πέμπτη του Στρασβούργου, αν δεν κάνω λάθος. Κάτι τέτοιο λέει ο πρόεδρος. 5 Νοεμβρίου, συζήτηση στην Ίντρε. Στην Ίντα 20 Νοεμβρίου 18 και ψηφίζουμε στην Ολομέλεια του Δεκεμβρίου. Να είστε έτοιμοι 8 Οκτωβρίου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Και να περάσουμε στο τελευταίο. Αποστολή της ΙΤΡΕΣ στην Νορβηγία, 7 με 9 Μαΐου 2018. Από ενημέρωση. Κύριε Βίρκουνεν, είναι μαζί μας σήμερα εδώ, αγαπητοί συνάδελφε. Σας ακούμε, αν και βλέπω εδώ ένα σωρό θέματα νομοθεσία στον τομέα της αγοράς ηλεκτρισμού και της πυρηνικής ενέργειας, λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, το μέλλον της βιομηχανίας φυσικού αερίου, δηληστήρια, καθαρές ενέργειες, απόδοση, διαχείριση απορριμμάτων. Μέσα σε τρεις μέρες θα καταφέρετε όλα αυτά. Μπράβο σας. Πώς τα καταφέρατε, κύριε μου. Ευχαριστώ. Εγώ μάλιστα έμεινα μόνο δύο ημέρες. Ο Σαλήν ήταν επικεφαλής τις τρεις τελευταίες μέρες. Είχαμε πραγματικά πάρα πολλά μπροστά μας να κάνουμε. Λοιπόν, πολύ γρήγορα. Γιατί βλέπω τον ευάριθμο πλήθος. Λάβατε την γραπτή έκθεση. Πάντως ήταν εξαιρετική επίσκεψη. Πολύ ενδιαφέρουσα για εμάς τους βουλευτές γιατί τρέχει και το Brexit τους τελευταίους μήνες. Η Νορβηγία είναι μία από τις χώρες που δεν είναι βεβαίως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά είναι ένας καλός εταίρος και για μας ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε από τους Νορβηγούς πώς βλέπουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση από εδώ και πέρα. Η αγορά ενέργεια είναι ένα πολύ ενδιαφέρον τομέα βεβαίω. Διότι ακριβώ η Νορβηγία δεν είναι μέλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όμως εφαρμόζουν σχεδόν όλη την ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον τομέα της ενέργεια, Τα θέματα τη ρήπανση, παράδειγμα, και έχουν συζητήσεις και στο κοινοβουλίο του ε, Κάποιοι λένε, μα γιατί αντιγράφεται την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εν πάση περιπτώσει, είναι σημαντικό η Νορβηγία να είναι μέρος της δικής μας ε, ηλεκτρικής αγοράς, αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μάλλον. Επίσης, συζητήσαμε τα θέματα ενεργειακή στρατηγική, διότι η Νορβηγία αξιοποιεί μόνο ανανεώσιμε πηγέ, πολλούν σε εμά και σε άλλου, όλο του το πετρέλαιο και όλο του το φυσικό αέριο δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα οι ίδιοι, να ξέρετε. Εμείς χρησιμοποιούμε τα δικά τους ορυκτά καύσιμα. Όταν α, μας τα πουλήσουν όλα, θα μας πουλήσουν και χώρους αποθήκευσης αποβλήτων. Πολύ έξυπνο από την πλευρά τους. Η μόνη πηγή ρήπαρση είναι η μεταφορά. Όμως σύντομα τα δύο τρίτα των οχημάτων τους θα είναι ηλεκτρικά, θα είναι ηλεκτροκίνητα. Και θα γίνουν λοιπόν ηγέτες και σε αυτόν τον τομέα. Πολύ ενδιαφέροντα όπως σας έλεγα για μας. Εστίασαμε φυσικά στην ενέργεια, όμως είχαμε και εξαιρετικές συζητήσεις επί θεμάτων έρευνας. Η Νορβηγία είναι σημαντικός εταίρος του Horizon 2020, διαφέρουσε επαφέ. Και επ' αυτού επισκεφθήκαμε θαλάσσιες πλωτέ δεξαμενές γεώτρηση. πήγαμε με ελικόπτερο και προσγειωθήκαμε εκεί και είδαμε ακριβώς τη δουλειά που γίνεται σε αυτές τις πλωτέ δεξαμένε, Μάλιστα κατεβήκαμε με, το ειδικό, τον ειδικό ελκυστήρα 300 μέτρα μέσα στη θάλασσα για να δούμε τις βάσεις αυτών των πλατφορών. Πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρον όπως φαντάζεστε. Μάθαμε πολλά για το πώς διαχειρίζονται την ενέργεια αλλά και την οικονομία τους αυτές τις τρεις ημέρες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε αγαπητή συνάδελφο για αυτήν την ενημέρωση. Και όπως θα είδατε υπήρχε και online αναμετάδοση και υπάρχει και η ομιλία σας ε, ε, στην ιστοσελίδα ε, της Επιτροπής μας. Οπότε είναι πολύ σημαντικό το ότι μας ενημερώσατε και ήταν πραγματικά σημαντική αυτή και πολύ ενδιαφέρουσα η επίσκεψη που κάνατε στην Ορβηγία. Ευχαριστούμε λοιπόν θερμά την κυρία Χαναβίργουνα ενός επικεφαλής αυτής της αντιπροσωπίας στην Ορβηγία. Και θα ήθελα να σας πω ότι οι επόμενες συνεδριάσεις μας είναι στις 8 Οκτωβρίου 3 έως 6.30 το απόγευμα και στις 9 Οκτωβρίου από τις 9 στις 12.30 και από τις 2.30 τις 6.30 το απόγευμα. Σε τρία, ας το πούμε έτσι, τμήματα η επόμενη συνεδρίασή μας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι από τα διάφορα. Εάν όχι, να περάσουμε στην επόμενη σε διάταξή μας και στο επόμενο σημείο της ημέρας διάταξης, δηλαδή η συνεδρίαση των συντονιστών. Οπότε κάποιοι από εσά μάλλον απαλλάσσεστε από τι ευθύνε σα και μπορείτε να εγκαταλείψετε την αίθουσα.